Νομίζω μπορούμε να αρχίσουμε με αυτή τη σημαντική προσέλευση των μελών. Beschlüsse der Αποφάσεις των συντονιστών. Της 31 Αυγούστου και οι σημερινές έχετε τα έγγραφα στα χέρια σας. Αν δεν διαφωνεί κανείς μέχρι το τέλος συνεδρίασης θα θεωρηθούν τα πρακτικά εγκεκριμένα. Οι αποφάσεις δηλαδή των συντονιστών ο κύριος Λούντγκρεν. Υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. Στο σημείο 3 γράφει ότι αποφάσισαν οι συντονιστές να δώσουν ε, τις ε, εκθέσεις εφαρμογή τους εισηγητές που ήταν εισηγητές για το θέμα αυτό αλλά χωρίς να γίνει ψηφοφορία ε, χωρίς να λέτε ποια είναι η μέθοδος αυτή, πώς αναθέσατε τις εκθέσεις. Εμείς δεν συμφωνούμε γιατί μας αποκλείουν εμάς ας πούμε από την ε, έκθεση γιατί δεν είχαμε στο παρελθόν ε, κάνει τις εκθέσεις. Και πώς πήρατε απόφαση. Απλώς το συζητήσατε. Ε, ζητούμε από τους εισηγητές να ξανασυνεδριάσουν και να βρουν ένα καλό τρόπο και μια ίση μεταχείριση γιατί δεν είναι σωστό να αποκλείονται μικρές ομάδες. Τι θα γίνει δηλαδή, δεν θα πάρουμε εμεί καμία έκθεση. Παρεξήγηση έγινε. Έγινε παρεξήγηση. Και γι' αυτό θα πρότεινα το εξή. Εφόσον είναι παρόν ο εισηγητής, αν είναι ξανά μέλος, το αναλαμβάνει. Άλλος, η ε, λόγω ομάδα του αρχικού εισηγητή θα αναλάβει την έκθεση. Εντάξει, αν το διαγράψουμε αυτό μπορεί να γίνει. Από ad hoc απόφαση, έτσι. Συμφωνείτε. Ωραία. Δεν υπάρχει άλλη διαφωνία για τα πρακτικά. Το συντονιστών είμαστε εντάξει. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Και προχωρούμε. Έλεγχος των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής. Παρουσίαση από τη Γενική Διεύθυνση MOVE. Το μέτρο ΚΔΕ κανονιστικής διαδικασίας ελέγχου σημαίνει αυτό, μεταξύ άλλων για την αεροπορία, συσκευές υποβρυχίου εντοπισμού, για τις θαλάσσιες μεταφορές, λιμενικές εγκαταστάσεις υποδοχής. Τέσσερις προτάσεις έχει κάνει πρόσφατα το Κοινοβούλιο ε, και είναι στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Μεταφορών. Το Κοινοβούλιο τώρα έχει τη δυνατότητα τα μέτρα αυτά να τα αξιολογήσει και να προβάλλει αντιστάσεις ή αντιρρήσεις εφόσον το θεωρεί απαραίτητο. Τα μέτρα με τα οποία θα ασχοληθούμε σήμερα αφορούν τις αεροπορικές και τις θαλάσσιες μεταφορές και μπορούν να ισχύσουν μόνο εφόσον το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο εντός τρίμηνης προθεσμίας δεν εκφράσει αντιρρήσεις ή επιφυλάξεις. Έχετε τα σχέδια από τις 26 Αυγούστου στο newsletter της Επιτροπολογίας μέχρι τις 27 Οκτωβρίου έχει το Κοινοβούλιο καιρό για να ε, διαφωνήσει βάσει ε, γνωμοδότησης και αιτιολογημένης της Επιτροπής Τραν. Θυμίζω ότι έχουμε ε, τρεις λόγους για να προβάλλουμε ενστάσεις κατά το μέτρο αυτό. Πρώτον, η πρόταση μέτρων υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεύτερον, δεν συνάδει με το στόχο ή και το περιεχόμενο του βασικού δικαίου δηλαδή της βασικής ε, νομικής πράξης και τρίτον αντιτίθεται στις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας. Όπως όλοι γνωρίζετε, στους τριμερείς ε, καταβάλουμε κάθε προσπάθεια στα νομοθετικά κείμενα να υπάρχει πάντα πολύ προσεκτική διατύπωση και το Κοινοβούλιο να αναφέρεται ότι έχει ε, τη δυνατότητα και την υποχρέωση ελέγχου. Τώρα λοιπόν έχουμε τέτοιες αρμοδιότητες που ανατέθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καλούμαστε να τις ελέγξουμε. Και είναι πολύ σημαντικό να τις μελετήσουμε σε βάθος και το χρόνο που χρειάζεται. Θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήρθε στο Κοινοβούλιο για να μας εξηγήσει όλα αυτά τα μέτρα. Τώρα καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, την Γενική Διεύθυνση ΜΟΥΒ, να μας παρουσιάσει τα εκτελεστικά μέτρα. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει σύντομα τέσσερα συνολικά τέτοια μέτρα και θα μιλήσει ο κύριος Φιλίπ Κορνέλης και στη συνέχεια η κυρία Κριστίν Μπέρκ. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Thank you, Mr. Um, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να ξεκινήσω με τα θέματα της αεροπλοείας. Λοιπόν, το πρώτο απ' όλα είναι ένα σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής να τροποποιηθεί ο κανονισμός 965 του 2012. Είναι ο κανονισμός OPS, όπως λέγεται με ακρονίμιο. Και αυτός ο κανονισμός έχει ως στόχο να εξετάσει μια σειρά, θεμάτων τα οποία έχουν προκύψει ε, σε αεροπορικά ατυχήματα. Έχουμε λοιπόν μάθει από διάφορα τέτοια ατυχήματα και έχουμε διαπιστώσει ότι μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο να εντοπίσει κανείς ε, το σκαρί του αεροσκάφους, κυρίως ε, όταν αυτό χάνεται ε, στο βυθό της θάλασσας. Πριν από κάποια χρόνια είχαμε την πτήση ε, της Air France ε, προς τη Βραζιλία. Εξαφανίστηκε ένα αεροσκάφος στην Ασία, επίσης πρόσφατα. Γι' αυτό λοιπόν θελήσαμε να εξάγουμε συμπεράσματα από αυτά τα δύο ατυχήματα. Και έτσι προτείνουμε μία νέα μέθοδο για να βελτιωθεί καταρχήν ο εντοπισμός του σκαριού του αεροσκάφους ε, και δεύτερον ο εντοπισμός του black box όπως λέγεται και επίσης ε, να μπορούμε να βρούμε μεθόδους, καλύτερες μεθόδους για να γνωρίζουν πάντα οι ε, αρμόδιοι που βρίσκεται η άτρακτος του αεροσκάφους ακόμα και αν ε, βρίσκεται το αεροσκάφος στον ωκεανό. Αυτή λοιπόν η μέθοδος εξυγχρονίζει καταρχήν τα black box που καταγράφουν τις φωνές. Είναι πολύ δύσκολο να το πιστέψετε αλλά μερικά αεροσκάφη εξακολουθούν για την μαγνητοφώνηση να χρησιμοποιούν τα παλιά κασετόφωνα. Άρα δηλαδή αυτά πρέπει να αντικατασταθούν. Επίσης ε, πρέπει να μπορούν αυτά τα μηχανήματα να ε, μαγνητοφωνούν 25 ώρες ε, της λειτουργίας. Παλιά ήταν μόνο 30 λεπτών ή 2 ώρων λόγω τεχνολογικών περιορισμών που δεν υπάρχουν όμως πλέον αυτή τη στιγμή. Αυτά για το black box. Τώρα για το τελευταίο αεροσκάφος προς την Ασία ουσιαστικά ε, μπορεί να προέκυψε η σύγκρουση αυτού του αεροσκάφου του ME370 e πολλές ώρες μετά την ε, αναστολή της καταγραφής. Προτείνουμε λοιπόν στο μέλλον να υπάρχουν βελτιωμένες συσκευές εντοπισμού υπό τον βυθό. Πρόκειται για πομπούς που εκπέμπουν ένα σήμα και έτσι οι αναζήτηση και διάσωση μπορεί πολύ πιο εύκολα να εντοπίσει την άτρακτο ε, για να μπορεί να γίνουν και οι σχετικές έρευνες. Σήμερα λοιπόν έχουν υπάρξει πολλές περιπτώσεις όπου αυτή η πομπή δεν είναι αρκετά ισχυρή και δεν μπορούν να λάβει, δεν μπορεί κανείς να λάβει το μήνυμά τους ε, από μακριά και τη στιγμή που ε, φτάνει κανείς ε, πλέον δεν υπάρχει τίποτα άλλο για να εντοπίσει το αεροσκάφος. Άρα δηλαδή χρειαζόμαστε ισχυρούς πομπούς που να λειτουργούν και στον βυθό της θάλασσας. Τώρα, ε, για την παρακολούθηση των αεροσκαφών. Εκεί προτείνουμε μία σειρά προδιαγραφών με βάση την απόδειση, έτσι ώστε στο μέλλον να είναι δυνατόν να εντοπιστούν τα αεροσκάφια όπου και αν βρίσκονται, ακόμα και στον ωκεανό. Δεν θα επιβάλλουμε μία συγκεκριμένη μέθοδο για να το κάνουμε αυτό. Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι στην αγορά. Πάντως ε, το βάρος βρίσκεται στον φορέα εκμετάλλευση για να πράξει όλα αυτά. Η ΙΚΑΟ, ο ΙΚΑΟ, ο οργανισμός ΙΚΑΟ συνεργάζεται και ο στόχος είναι να υπάρχει συντονισμός με τους διεθνείς κανόνες, κάτι που πάντα προσπαθούμε να κάνουμε όταν μιλάμε για τεχνικές προδιαγραφές ε, των αεροσκαφών. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία του πρώτου φακέλου. Αν θέλετε να συνεχίσω και για τα υπόλοιπα, Τώρα, ο δεύτερος και ο τρίτος φάκελος αφορούν πάλι το ίδιο θέμα που είναι το επίπεδο της συγχωρήπανσης για τα αεροσκάφη. Ε, υπάρχουν δύο κείμενα και αφενός τροποποιούνται οι βασικοί κανονισμοί ασφάλειας που είναι κανονισμοί του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου και κατά δεύτερον τροποποιούμε μία σειρά εφαρμοστικών κανονισμών που έχουν εγκριθεί. Ε, το αντικείμενο είναι πάντα το ίδιο, δηλαδή να υπάρχει ένα νέο επίπεδο χορύπανση για τα μελλοντικά αεροσκάφη για το μελλοντικό τύπο αεροσκαφών. Όπως τα ξέρετε, στο πλαίσιο του ΙΚΑΟ έχουμε ήδη δουλέψει πολλά χρόνια σχετικά με αυτό το επίπεδο η χορύπανσης, έτσι ώστε οι κατασκευαστικές εταιρείες αεροσκαφών να προχωρούν όλο και πιο πολύ όσο το επιτρέπει η τεχνολογία για να δώσουν το μέγιστο που μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία για να περιοριστεί η χορύπανση. Άρα δηλαδή αυτή τη φορά έχουμε χαμηλότερα όρια, ανώτατα όρια για τα μελλοντικά αεροσκάφη και με την πάροδο του χρόνου θα είμαστε όλο και πιο αυστηροί. Δηλαδή προτείνουμε νέες προδιαγραφές που βασίζονται στις ε, προηγούμενες για να είμαστε, όπως σας είπα, όλο και πιο αυστηροί για αεροσκάφη τα οποία βγαίνουν ή θα βγουν στο μέλλον στην αγορά. Όλα αυτά βασίζονται απόλυτα σε δουλειά που κάνει ο ΙΚΑΟ και εμείς βεβαίως έχουμε συμβάλει τα μάλα ως Ευρώπη. Αν θέλετε κατά κάποιον τρόπο ήμασταν ε, η κινητήρια δύναμη όλων αυτών διότι ο θόρυβος και η χορύπανση είναι πολύ μεγάλο θέμα για μια πυκνοκατοικημένη περιοχή όπως είναι η Ευρώπη και γι' αυτό πιέζουμε όσο μπορούμε. Έτσι λοιπόν το Συμβούλιο του ΙΚΑΟ ενέκρινε τροπολογίες ε, στο παράρτημα 63 που είναι οι σχετικοί κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος του ΙΚΑΟ. Ε, το, στις 14 Μαρτίου τίου λήφθη απόφαση και εμείς είπαμε ότι οι κανονισμοί αυτοί θα πρέπει να ενταχθούν στο δικό μας το νομοθετικό πλαίσιο. Κατ' ουσίαν δεν έχουμε καμία άλλη δυνατότητα γιατί και στους δικούς μας κανονισμούς προβλέπεται να εφαρμόζονται ακριβώς οι ίδιοι κανονισμοί που εφαρμόζει και ο ΙΚΑΟ για το περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, οι νέες προδιαγραφές ε, ε, αναφέρονται σε 7 δεσιμπέλ τα νέα στάνταρ οι νέες προδιαγραφές ε, θα εφαρμόζονται στα νέα τύπη αεροσκαφών, τα JET και θα υποβληθούν αυτές οι προδιαγραφές για ε, πιστοποίηση από το 2014. Θα ε, αφορούν τα μεγάλα αεροσκάφη 55 τόνων και μετά το 2020 θα έχουμε, τα, θα ισχύουν για jet αεροσκάφη κάτω των 55 και για τα ελικοφόρα που επίσης για το οποίο προβλέπεται ένα συγκεκριμένο βάρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέει ο Πρόεδρος, δεν ξέρω αν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια επ' αυτού. Ο κύριος Κούν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να πω όλα αυτά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα Ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις πληροφορίες ε, σχετικά με τα νέα μέτρα. Και αυτά, από ό,τι φαίνεται, προέκυψαν λόγω των σοβαρών αεροπορικών ατυχημάτων των τελευταίων ετών. Τώρα λοιπόν τα αεροσκάφη θα είναι εξοπλισμένα με καλύτερους ασυρμάτους, όχι μόνο με τα black box και με το κουτί το, της μαγνητοσκόπησης, μαγνητοφώνησης με συγχωρείτε ήχου, έτσι ώστε ε, τα αεροσκάφη αν συντριβούν μετά από οξύτατη σύγκρουση να μπορεί κανείς ε, και μετά από 24 ώρες ε, να παρακολουθήσει τι ακριβώς έχει διαδραματιστεί. Όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα. Επίσης είναι σημαντικό να υπάρχει συντονισμός με τον ΙΚΑΟ και δηλαδή με τον Διεθνή Οργανισμό Αεροπολίας και με τον Ευρωπαϊκό. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ανατολική Ουκρανία και ε, υπάρχει υποψία για κατάρριψη επιβατικού αεροσκάφους σε αυτό τον εναέριο χώρο. Η σύγχυση που προέκυψε με το να κλείσει ή όχι ε, ο ενάριος χώρος μέχρι 11.000 ε, πόδια, αυτό... Μέτρα. μέτρα, μέτρα με συγχωρείτε. Όμως ακόμα και αν έγινε αυτό θα, μπορούσαν, ε, θα μπορούσε να έχει πληγεί το αεροπλάνο και μέχρι 30.000 μέτρα. Υπήρξαν κάποια αεροσκάφη της British Airways που δεν περνούσαν μέσα από αυτόν τον αέριο χώρο, όμως ε, τα αεροσκάφη της Malaysian Airlines διέσχιζαν αυτό το χώρο. Εκεί λοιπόν θέλω να ρωτήσω τι έγινε ε, προβλέπονται συγκεκριμένα μέτρα ε, κατεξοδότηση, πράξη ή οτιδήποτε το σχετικό. Ο κύριος Λούντγκριν. Τα περισσότερα που θέλω να ρωτήσω τα ρώτησαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι, οπότε δεν θα ρωτήσω τίποτε. Ο κύριος Γκόλνης. Ευχαριστώ πολύ. Τα μέτρα που προτάθηκαν μου φαίνονται πολύ λογικά εκ πρώτης όψεως, όμως θέλω να, να θέσω το εξή ερώτημα. Ποια είναι η σχέση με ε, τα πρότυπα ε, που διατυπώνονται από τον ΙΚΑΟ, από το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, Υποθέτω ότι οι προδιαγραφές ε, θα είναι αυστηρότητες, αυστηρότερες από του ΙΚΑΟ, γιατί διαφορετικά δεν υπάρχει λόγος ύπαρξής τους και βέβαια αυτό οδηγεί σε άλλα ερωτήματα συγκεκριμένα όσον αφορά ας πούμε τις προδιαγραφές που αφορούν ε, τα επίπεδα του ήχου, την ύπανση. Αυτοί οι κανόνες θα ισχύουν μόνο για τους Ευρωπαίους κατασκευαστές ή θα επιβληθούν ε, για όλα τα αεροσκάφη που θα κάνουν υπερπτήση ε, στην Ευρώπη για να το πω αλλιώς, πώς μπορούμε να επιβάλλουμε τις προδιαγραφές αυτές εκτός Ευρώπης και αν δεν το καταφέρουμε αυτό, μήπως θα δημιουργηθεί έτσι αθέμητος ανταγωνισμός ε, από κατασκευαστές ε, αεροσκαφών ε, που δεν θα είναι Ευρωπαίοι και που δεν θα χρειάζεται να ακολουθήσουν ε, τις προδιαγραφές αυτές που θα ισχύουν για την Ευρώπη. Δεν βλέπω να ζητά κανείς άλλο το λόγο. Παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ. Το πρώτο ερώτημα για την Ανατολική Ουκρανία. Καταρχάς πρέπει να πω ότι αυτό είναι εκτός ε, του ε, πεδίου εφαρμογής ε, του κανονισμού που εξετάζεται τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρ' όλα αυτό, αυτά να πω ότι έχουν γίνει προσπάθειες από το MS, το MS17 την πτήση MS-17, να δούμε ακριβώς τι συνέβη διότι δεδομένη της διεθνής ε, νομοθεσία, νομοθεσίας, ε, οι ίδιες οι αεροπορικές εταιρείες αποφασίζουν ε, ποιο δρομολόγιο θα ακολουθήσουν. Ο ΙΚΑΟ ανταλλάσσει πληροφορίες, ζητά, ζητά από τις αεροπορικές εταιρείες να ανταλλάσσουν καλύτερα Ε, μέσω του Νόταμ τις πληροφορίες ε, ε, μεταξύ των αεροπορικών εταιριών πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά και στο πλαίσιο αυτό η ΕΑΖΑ και που πρέπει παρεπιπτόντος να την ευχαριστήσω γιατί προετοιμάζει όλους αυτούς τους κανονισμούς για μας. Κάτι ακόμη λοιπόν που έχει κάνει η ΕΑΖΑ είναι να δημοσιοποιήσει περισσότερο ε, τις ε, πληροφορίες για ένα αέριο χώρο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και συστάσεις προς τις αεροπορικές εταιρείες. Ε, αυτά μπορώ να σας πω που σας είπα είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού που εξετάζουμε σήμερα. Όσον αφορά τώρα το επίπεδο της ηχορύπανσης και τις σχετικές προδιαγραφές κατά πόσο είμαστε εμείς αυστηρότεροι από τον ΙΚΑΟ. Όχι, δεν είμαστε. Ε, η υφιστάμενη νομοθεσία ε, η οποία μας ε, διέπει, μας επιτρέπει να αντιγράψουμε επακριβώς προδιαγραφές του ΙΚΑΟ, τίποτε παραπάνω και τίποτε λιγότερο. Αυτό βάσει του κανονισμού 216 του 2008. Είναι σημαντικό να μεταγράψουμε αυτές τις προδιαγραφές στη δική μας νομοθεσία, γιατί δεν έχουν άμεση ε, δεν, δεν είναι άμεσα δεσμευτικές ε, μέσω του ΙΚΑΟ. Πρέπει να καταστούν ε, δεσμευτικές για τους Ευρωπαίους κατασκευαστές μέσω της εφαρμογής αυτών των κανονισμών. Ε, τα, οι προδιαγραφέ αυτέ αφορούν του κατασκευαστέ, αλλά όχι του χειριστέ των αεροσκαφών και αυτό σημαίνει ότι κάθε νέο αεροσκάφο που θα τοποθετείται στην αγορά μετά από την ε, ημερομηνία που αναφέρεται εδώ πρέπει να συνάδουν με τι προδιαγραφέ συγχωρήπανση. Δεν υπάρχουν τόσοι κατα, κατασκευαστές ε, μεγάλων αεροσκαφών στον κόσμο. Έχουμε την Airbus εμεί βέβαια που θα δεσμεύεται από αυτές τις προδιαγραφέ. και είναι και άλλε εταιρείε από τον Καναδά Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες και, ε, και τη Βραζιλία. Όμως για την ώρα ε, αυτές είναι οι μόνες χώρες ε, που κατασκευάζουν τέτοιου μεγέθους αεροσκάφη και και αυτές δεσμεύονται από τις προδιαγραφές αυτές του ΙΚΑΟ για τα σκάφη για τα οποία είναι υπεύθυνα. Οπότε δεν βλέπω κανένα πρόβλημα με την εφαρμογή χαμηλότερων προδιαγραφών. Ευχαριστώ. Ο κύριο Σκούν έχει μια συμπληρωματική διευκρινιστική ερώτηση, μικρή. Για τα όρια που θα πρέπει να τεθούν ε, ανώτατε τιμέ για την ηχορύπαση και το θόρυβο από το 2018. Πάνω από 50 τόνους συνολικό ε, βάρος των αεροσκαφών Κοιτάξτε, ποιος κάνει θόρυβο, οι τουρμπίνε Και οι εταιρείε που κατασκευάζουν τουρμπίνε, μεταξύ άλλων η Rolls Royce είναι μια πολύ μεγάλη και γνωστή. Και είναι και ένας από τους παγκόσμιου ηγέτε. Αν ορίζουμε τέτοιες τιμές και στη συμφωνία με τον ΙΚΑΟ, τα αποτέλεσματα της έρευνας και της ανάπτυξης ε, δεν θα πρέπει να είναι τέτοια που να έχουμε μια τέλεια καύση με μείωση του θορύβου από το 2018 ήδη από τότε στις τουρβίνες που να μπορούν να κυκλοφορούν στην αγορά. Οι κινητήρε αυτοί θα πρέπει να είναι ρεαλιστικά, αλλιώ μπορούμε να βάζουμε οριακέ τιμέ για το θόρυβο που δεν ε, είναι ε, τεχνολογικά εφικτά. Όλα τα αεροπλάνα, δηλαδή τα αεροσκάφια που θα κυκλοφορούν και θα παράγονται από το 2018 και μετά, πάνω από τους 55 τόνους ας πούμε συνολικό βάρος, θα πρέπει να έχουν ένα τέτοιο όριο δεσιμπέλ και από το 2021 και πιο κάτω. Και μιλώ όχι μόνο για τα αεριοθούμενα, αλλά και για τα ελικοφόρα. Γιατί εκεί είναι και άλλοι ε, οι κατασκευαστές, είναι η Airbus, ε, Lockheed, ε, Boeing κτλ. Τεχνικά είμαστε καλυμμένοι, το έχετε ψάξει αυτό. Σύντομη απάντηση. Ναι κύριε Κούν. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή είναι η, η δυσκολία τη διαδικασία και αυτό κάνουν οι εμπειρογνώμονε όταν προετοιμάζουν τις προδιαγραφές ε, ε, ε, στον ΙΚΑ. Όπως είπα, είμαστε πολύ δραστήριοι με τη βοήθεια της ΕΑΖΑ και των μηχανικών της από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσουν τι προδιαγραφέ σε τέτοιο επίπεδο ώστε να είναι τεχνικώ εφικτέ, αλλά να είναι όσο το δυνατόν πιο φιλόδοξε, να πιέσουν, να ε, πιέσουν ε, τον τομέα να εξελιχθεί, χωρίς βέβαια να επιβάλλονται προδιαγραφές ε, οι οποίες θα παρεμποδίσουν το σχεδιασμό νέων αεροσκαφών. Εν ολίγης, τα πιστοποιητικά ηχορύπανσης ισχύουν, πρέπει να εκδοθούν και για τα Boeing και για τα Airbus. Βέβαια, αυτός είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας, δεν είναι το πιο βασικό, αλλά είναι ένας καθοριστικός παράγοντας. Μια που αναφέρθηκε η Rolls Royce. Θυμάμαι μια συζήτηση πριν από 40 χρόνια με συνδικαλιστές που μου είπανε ότι η Rolls Royce φτιάχνει αυτοκίνητα που είναι τόσο θόρυβα που δεν τα ακούς στο δρόμο. Αλλά εκείνοι που κατασκευάζουν τους κινητήρες στα εργοστάσια, οι άνθρωποι καταστρέφονται από το θόρυβο. Δηλαδή, ε, το τι είναι δυνατόν ε, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα από αυτά που συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση και πάμε στην επόμενη της κυρίας Κριστίν Μπέρκ. Ευχαρίστως. Ε, πηγαίνουμε από τον αέρα στη θάλασσα και περνάμε σε ένα περιβαλλοντικό θέμα. Αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η τροποποίηση ενός παραρτήματος ε, στην υφιστάμενη οδηγία του 2000 ε, για τις, τις καταστάσεις λιμενικής υποδοχής και για τη χρήση, για την επεξεργασία των λιμάτων και των αποβλήτων. Ε, υπάρχουν ε, πληροφορίες τις οποίες πρέπει ε, ένας πλοίαρχος να δώσει όταν μπαίνει σε ένα λιμένα. Βάσει της οδηγίας δεν επιτρέπεται τα απόβλητα των πλοίων να απορρίπτονται στη θάλασσα, αλλά πρέπει να εκφορτώνονται σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις υποδοχής, τις οποίες πρέπει να παρέχουν οι λιμένες. Ε, στη διεθνή νομοθεσία ε, είναι ε, πολύ, είναι, είναι, με, πολύ ευρύς αυτός ο τομέας. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες στο πλαίσιο της Διεθνούς Οργάνωσης Ναυτιλίας και MAPL είναι η σύμβαση που ισχύει. Ακούσαμε κάποια πράγματα για τον ΙΚΑΟ, είναι παρόμοια η κατάσταση θέλουμε μια ε, πιο λεπτομερή κατηγοριοποίηση των ε, προκαλούμενων από τα ε, πλοία αποβλήτων από αυτήν που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην οδηγία. Και επομένως η ιδέα είναι να ενημερώσουμε τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στα ευρωπαϊκά λιμάνια και να ευθυγραμμιστούν με τις διεθνείς, με τις διεθνείς απαιτήσεις ώστε να είναι ισότιμο το πεδίο διεθνώς. Όσον αφορά την παροχή των πληροφοριών αυτών ε, που πρέπει να παρέχει ο πλήρχος δηλαδή ε, ποιος είναι ο όγκος των αποβλήτων ε, και ε, πόσο αποθηκευτικός χώρος θα έπρεπε να υπάρχει σε ένα πλοίο για να μπορεί να μην ε, έχει την υποχρέωση να εκφορτώσει τα απόβλητα μέχρι να πάει στον επόμενο λιμένα. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε κατά πόσο υπάρχει αποθηκευτικός χώρος για να είμαστε βέβαιοι ότι δεν απορρίπτονται παρανόμως στη θάλασσα τέτοιου είδους πληροφορίες πρέπει να παρέχονται ηλεκτρονικώς, ε, κάτι που δεν είχε προβλεφθεί το 2000 ε, όταν άρχισε να ισχύει η οδηγία. Όμως τώρα υπάρχουν ηλεκτρονικά συστήματα αναφορών ε, που θα δώσουν την δυνατότητα να συλλέγονται αυτές οι πληροφορίες και να διαχέονται μεταξύ των λιμενικών αρχών ηλεκτρονικός. Πιστεύουμε ότι η κατάσταση με, την ε, τροποποίηση της οδηγίας αυτής είναι επικερδής για όλους, ότι είναι ευκολότερο για τις αρχές τήρησης του νόμου να δουν κατά πόσο κάποιο ε, ε, σκάφος πρέπει να εκφορτώσει τα απόβλητά του ή να συνεχίσει. Σε διαφορετική περίπτωση θα απορριφθούν στη θάλασσα, επομένως από περιβαλλοντικής απόψεως κερδίζουμε κάτι και είναι πολύ καλύτερο και από απόψεως ανταλλαγής πληροφοριών γιατί το να, ε, στέλ, να αποστέλλονται οι πληροφορίες ηλεκτρονικώς σημαίνει ότι ε, δεν χρειάζεται να γίνει διαδικασία στον πρώτο λιμένα ε, εφόσον έχει ήδη διαπιστωθεί ότι μπορεί να συνεχίσει το ταξίδι του, το σκάφος μέχρι τον επόμενο λιμένα και να κάνει εκεί την εκφόρτωση. Η εμπειρογνώμονάς μας ε, μπορεί να σας ε, κάνει και μια πιο λεπτομερή παρουσίαση, αν θέλετε. Ευχαριστώ πολύ. Ερωτήσεις, έχετε σχόλια. Ο Βιμ Βαντεκάμπ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Κατανοώ ότι όλοι θέλουμε οι θάλασσές μας και τα πελάγη μας να είναι καθαρά και αυτό θέλω να ρωτήσω. Ε, μόνο για τη θάλασσα μιλάμε για εσωτερική ναυσιπλοεία, για τα ποτάμια, για τις εσωτερικές πρωτοέσοδους επίσης. Και δεύτερη ερώτηση. Οι λιμένες θα είναι υποχρεωμένοι να έχουν μια χωρητικότητα, μια δυνατότητα να υποδέχονται όλα αυτά τα απόβλητα. Διότι καλό είναι να λέτε στα καράβια να τα ρίχνουν αυτά στα λιμάνια, αλλά αν δεν έχουν τη δυνατότητα απορρόφησης οι λιμένες, τι γίνεται. Γιατί έχουμε και καλά λιμάνια και λιγότερο καλά και μεγάλο ανταγωνισμό μεταξύ των λιμένων. Μήπως μπορείτε να μου το απαντήσετε αυτό, αυτά τα δύο ερωτήματα. Ευχαριστώ πολύ. Gibt's weitere Ο Κούν. Κοιτάξτε, είναι γνωστό ότι στα μεγάλα εμπορικά σκάφη υπάρχουν εγκαταστάσεις καύσης αποβλήτων, καυσι, αποβλήτων. Το τι θα κάνουμε λοιπόν, το κατά πόσον ε, θα μπορούμε τις αποθήκες για τα απόβλητα, ε, το μέγεθος μάλλον αυτών των αποθηκών, να το προσαρμόζουμε στη διάρκεια πλεύσεις των σκαφών. Δεν ξέρω, έχετε προβληματιστεί επ' αυτού. Γιατί νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να τηρείται από την αρμόδια αρχή ελέγχου του λιμένος. Δηλαδή, δεν θα ελέγχονται μόνο τα εμπορικά σκάφη, τα φορτηγά, το κατά πόσον πράγματι τηρούν όλες τις προδιαγραφές σχετικά με το, ε, τους εργαζόμενους, ε, τους επιβάτες, οτιδήποτε, αλλά και το μέγεθος της αποθήκης αποβλήτων. Θα πρέπει να ελέγχεται και αυτό. Και κατά πόσον και το λιμάνι έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης. Αυτό το συγκεκριμένο ποιος θα το ελέγχει, πρόεδρος. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, ε, θα κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Κοιτάξτε, οι μεγαλύτερες εγκαταστάσεις ε, καύσης ε, αποβλήτων είναι τα υπεροκεάνια, διότι αυτά χρησιμοποιούν μαζούτ και το μαζούτ είναι προϊόν της καύσης. Άρα δηλαδή αυτό που παίζει ρόλο είναι ότι αν αναγκαστούν τα υπεροκειάνια, τα μεγάλα φορτηγά να εγκαταστήσουν άλλες μονάδες, τότε καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχουν ε, και μεγαλύτερες εκπομπές. Εκτός αν βάλουν φίλτρα. Αυτό όμως κοστίζει και θα διαμαρτυρηθούν. Γιατί τα καύσιμα των σκαφών είναι πολύ φτηνά, πάρα πολύ φτηνά. Ερωτώ λοιπόν, θα κάνετε κάτι σχετικά με αυτό. Βεβαίως και είναι σημαντικά τα απόβλητα να μην ε, κλείονται στη θάλασσα, αλλά και αυτό που σας ρώτησα εγώ και αυτό με ενδιαφέρει. Κοιτάξτε, να εξετάσω ερωτήσεις μία προς μία με τη σειρά που ετέθησα. Να καταστήσω απόλυτα σαφές ότι αυτή η οδηγία δεν αφορά την εσωτερική ναυσιπλοεία. Μιλάμε για θαλάσσιους λιμένες και όπως έχει ήδη αναφερθεί από τους συναδέλφους, οι λιμένες είναι υποχρεωμένοι να έχουν την υποδομή για να δέχονται τα απόβλητα τα οποία έχουν προκληθεί από την πλεύση των σκαφών. Υπάρχει βέβαια μία προϋπόθεση ότι όλα αυτά θα πρέπει να είναι και λογικά και πρακτικά εφαρμόσιμα. Γιατί επειδή υπάρχουν πάρα πολλά σκάφη, με συγχωρείτε λιμάνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν και μικρές αθλητικές μαρίνες. Δεν μπορεί τώρα κανείς να περιμένει αυτή η υποδομή να προσφέρεται και στο Ρότερνταμ και σε ένα μικρό ελληνικό νησί. Εξαρτάται πάλι και από την ε, κίνηση που έχει ένα λιμάνι. Δεν μπορεί κανείς να περιμένει ένα λιμάνι το οποίο επισκέπτεται μια φορά το χρόνο ένα αν θέλετε σκάφος, ίσως ένα κρουαζιερόπλιο, να έχει την ίδια υποδομή όπως ένας άλλος λιμένας που δέχεται τακτικά σκάφη. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να το γνωρίζουν οι εποπτικές αρχές Μπορεί να υπάρχει έλεγχος, αλλά όχι υποχρεωτικά. Αυτό είναι στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών. Μην ξεχνάτε επίσης ότι σε τέτοιου είδου ελέγχους, ε, μάλλον αυτοί οι έλεγχοι αφορούν ε, τα ε, σκάφη με ξένες σημαίες. Οι έλεγχοι θα γίνονται αλλά όχι όπως σας είπα υποχρεωτικά. Και κάτι το οποίο είναι σημαντικό είναι το εξής όταν ε, γίνεται ο έλεγχος δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν τα πάντα όλοι υποδοχείς ε, που υπάρχουν ας πούμε ε, για τα κατάλοιπα των καψίμων. Δεν γίνεται αυτό σε κάθε έλεγχο. Ανάλογα με το σχεδιασμό του σκάφους από εκεί ε, προβλέπεται και πόσο μεγάλη θα είναι η δυνατότητα αποθήκευσης. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι τα σκάφη μετακινούνται από λιμένα σε λιμένα. Ε, γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να υπάρχει ένα ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο θα βοηθάει τις αρμόδιες αρχές ε, και κάποιον άλλον που εκπροσωπεί αν θέλετε το Υπουργείο Περιβάλλοντος να μπορεί πριν ακόμα το σκάφος μπει στο λιμάνι να ελέγξει ηλεκτρονικά κατά πόσον υπάρχει ακόμα κάποιο περιθώριο αποθήκευσης αποβλήτων. Αν όχι, τότε θα πρέπει να το έχει κατά νου γιατί από τη διαδρομή που είναι σαφής, καθίσταται σαφές ότι το αεροσκάφι, το, το θα μπορεί να πάει στο επόμενο λιμάνι αν δεν αδειάσει κάποια απόβλητα στη θάλασσα. Επίσης ε, υπάρχουν όπως σας είπα αυτές οι υποδοχείς ε, καυσίμων ε, πάνω στα σκάφη Το είπε. στα κουρασγερόπλια. Επίσης, αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτοί, αυτές οι εγκαταστάσεις κάψης μπορεί να είναι πολύ τοξικές, γιατί χρησιμοποιούν ή εκεί υπάρχουν οξέα που δεν βρίσκονται στα φυσιολογικά απόβλητα σκουπίδια. Άρα δηλαδή τώρα αλλάζει εδώ η κατηγοριοποίηση των αποβλήτων. Ως εκ τούτου τα μεγάλα λιμάνια θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι θα μπορούν να δέχονται όλο και περισσότερα τοξικά απόβλητα καθότι όπως σας είπα εφόσον εγκαθίσταται αυτή η τεχνολογία καύσης ε, προβλέπεται και αυτή η κατηγορία των αποβλήτων στα μεγάλα ε, επιβατηγά πλοία. Επίσης, αυτό που έχει σημασία είναι τα λιμάνια να προσφέρουν κάποιες δυνατότητες. Ε, τα χρεώνουν τους ε, φορείς εκμετάλλευσης των σκαφών, θα δίνουν κίνητρα έτσι ώστε να μην προκαλούνται τόσα πολλά απόβλητα από τα σκάφη. Άρα δηλαδή, εάν ληφθούν μέτρα ώστε να περιορίζονται τα απόβλητα ήδη πάνω στο σκάφος, τότε αυτό είναι κάτι που θα πρέπει οι λιμένες να το λαμβάνουν υπόψη τους όταν χρεώνουν τα τέλη για τις υπηρεσίες που προσφέρουν, δηλαδή για την υποδοχή των αποβλήτων. Τώρα, σε αυτό που είπατε, κάνατε μία ερώτηση. Είπατε ότι τα σκάφη, τα μεγάλα ποντοπόρα σκάφη, σήμερα τα κατάλοιπα των βρώμικων καψίμων, όχι μόνο τα εμπορευματοκιβώτα ε, φορτηγά, αλλά και τα κουρασγερόπλια, Και αυτά ε, έχουν αυτά τα κατάλοιπα αλλά εγώ θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια σχετική νομοθεσία για να βελτιωθεί η σύνθεση, κυρίως η περιεκτικότητα θείου. Άρα δηλαδή αυτά τα σκάφη καλούνται να χρησιμοποιούν πιο ελαφριά καύσιμα που δεν είναι τόσο βρώμικα ή χρησιμοποιούν περίφημες τα scrubbers, τις πλύντρες. Ε, νομίζω ότι θέλω να, πω, να επισημάνω το εξής. Ενώ αυτό το μέτρο προτείνεται κυρίως σε σχέση με την κατηγοριοποίηση των αποβλήτων που προτείνεται σε διεθνές επίπεδο, πάλι σε διεθνές επίπεδο έχει σαχθεί ε, και μία νέα κατηγορία καψίμων, είναι τα απόβλητα ακριβώς από αυτές τις πλύντρες. και αυτό προβλέπεται στη σύμβαση Μάρπολ. Όπως ε, είπατε κι εσείς, ε, στην αρχή μόλις ξεκινήσαμε υπάρχει και μια σωστά ε, οριζόμενη παράμετρος για το τι ακριβώς μπορεί να κάνει η Κομισιόν και επίσης και να προτείνει με τέτοιου είδους μέτρα. Αν τελικά προτείνουμε με αυτή τη διαδικασία μια νέα μορφή η κατηγορία αποβλήτων αυτή θα ξεπεράσει το πεδίο εφαρμογής οδηγίας γιατί αυτή ανάγεται στο 2000 η οδηγία. Και τότε ε, λοιπόν τα ε, τοξικά τα απόβλητα που προκύπτουν από τις πλύντρες όπως είπαμε δεν υπήρχαν, κανείς δεν τα είχε σκεφτεί, πλυντρίδες πολύ σωστά. Έτσι λοιπόν ε, είμαστε πλέον αναγκασμένοι να δούμε να αξιολογήσουμε την ε, λειτουργία, την εφαρμογή της οδηγίας και κατά πάσα πιθανότητα το 2017 θα προτείνουμε να αναθεωρηθεί ολόκληρη η οδηγία και τότε θα πρέπει να επεκτείνουμε και το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για να μπορούμε να συμπεριλάβουμε και αυτή τη νέα κατηγορία ε, αποβλήτων που δεν καλύπτεται αυτή τη στιγμή. Ε, θα ήθελα λοιπόν να σας διαβεβαιώσω για το εξής. Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι συμβαλόμενα μέρη της Συμφωνίας Μάρπολ και η αναθεώρηση της Συμφωνίας Μάρπολ σε σχέση με τις κατηγορίες, την κατηγοριοποίηση των αποβλήτων, αυτή ετέθησε ισχύ η Συμφωνία το 2013. Άρα δηλαδή στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει τα κράτη-μέλη έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις αυτή για την οποία συζητάμε σίγουρα, αλλά ακόμα δεν μπορούμε να επιβάλλουμε κάτι μέσα από οδηγία, γιατί αν η Κομισιόν πρότεινε να εισαχθεί αυτή η νέα κατηγορία αποβλήτων, κάτι που όμως δεν είχε συμφωνηθεί μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου το τότε ε, θα αφήναμε ένα τεράστιο περιθώριο ελιγμών. Αυτά είχα να σας πω και σας ευχαριστώ πολύ. Χωρίς μικρόφωνο Πρόεδρος, το λόγο ο κύριο Κούν. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που συζητάμε τώρα και για ε, τις εφαρμοστικές διατάξεις και να τις συζητούμε και σε σχέση, σε μία με την άλλη. Πέρσι και προ, ε, ε, πέρσι είχαμε συζητήσει έτσι πάρα πολύ θερμά για τα θέματα του θείου από την 1η του 2015 θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες περιφέρειες που να είναι ελεύθερες εκπομπών θείου στη Βαλτική θάλασσα, στη Βόρεια θάλασσα μέχρι την Ανατολική Μάχη αλλά και την Νορβηγία ε, που βρέχεται από τη θάλασσα και ε, από την άλλη μεριά είναι ε, στην Σκοτία. Ε, όχι, λιγότερο από 0,1% θείο επιτρέπεται να είστε στη δεξαμενή και μέχρι το 2020 σε ένα δεξαμενόπλιο αυτό θα πρέπει να αφορά όλα τα ύδατα. Αυτό δεν είναι ποιότητα ντίζελ και σωστά είπε ο πρόεδρος ότι αν δούμε τα υπολείμματα που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, ε, ε, πουθενά αλλού εκτός από διάφορες τουρμπίνες είναι ο μεγαλύτερος βαθμός ρήπανσης. Και αυτό για τα ποντοπόρα επιτρέπεται, 3,5% θείο και στις σε ελεγχόμενες περιοχές, αν θυμάμαι καλά, είναι 0,1% και αυτό έχει να κάνει με ε, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα κτλ. κτλ. Και θα με ενδιέφερε να μάθω πώς βρίσκεται η κατάσταση των διαπραγματεύσεων μεταξύ κρατών μελών και Μάρπολ, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι συμβαλόμενο μέρος στη Μάρπολ ε, τα αποτελέσματα μόνο της οδηγίας για το θείο θα πρέπει να τα εφαρμόσουμε. Από το 2020 αυτό θα το έχουμε πετύχει, να είναι 1% μόνο στη δεξαμενή ε, και αυτό το μαζούτ, το υπόλοιμα που ε, αν βγάλει την ελαφρία βενζίνη και το ντίζελ και έχει καεί όλο αυτό το καύσιμο και μένει αυτό το περίτομα για να το πω έτσι, ε, το καίνε τα καράβια. Ε, κανονικά αυτό άμα πάλι σε ένα φτιάρι, το, το φτιάρι ε, κολλάει μέσα και ε, για να το βγάλεις θα πρέπει να θερμανθεί και να μπει σε ένα μεγάλο καυστήρα, ελεύητα και σε μια εγκατάσταση που θα πρέπει να το υγροποιήσουν για να καεί. καταλαβαίνετε ότι αυτή η κατάσταση... θα πρέπει να εφαρμοστεί παγκοσμίω στις ε, Μαρπόλ. Οι Αμερικανοί βάλαν ζώνη 200 ναυτικά μίλια. Εμείς μόνο στο βορρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Θείο, αλλά θα πρέπει να επεκταθεί και στα υπόλοιπα ύδατα και στη Μεσόγειο και αλλού. Και θα με διέφερε πώς ε, κυμαίνονται οι συζητήσεις αυτό τον καιρό και οι διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Και τώρα με πολύ μεγάλη περιέργεια περιμένουμε την απάντηση. η κατάσταση των πραγμάτων έχει ως εξής. Αυτές οι περιοχές για την ενελχόμενη εκπομπή θείου ε, στην Βόρεια Αμερική έχουν να κάνουν και με τα οξύδια του αζότου, όχι μόνο με το θείο. Ενώ εμείς στην Ευρώπη με την οδηγία έχουμε ορίσει ε, όρια ε, και έχουν τεθεί σε ισχύ αυτές οι οδηγίες. Αλλά παγκοσμίω αυτό δεν συμβαίνει έτσι. Εάν πάτε στο Παγκόσμιο Οργανισμό Ναυσιπλοείας, ΑΕΜΟ, μόνο η Βόρειο Αμερική και η Ευρώπη έχουν αυτές τις αυστηρές προδιαγραφές από όλο τον κόσμο. Η σημερινή συζήτηση όμως δεν αφορά τις εκπομπές ε, που βγαίνουν από το φουγάρο, αλλά γιατί έχουμε περιορισμούς για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και η κατάσταση έχει ως εξής. Ε, ορισμένοι πλειοκτήτες αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν ε, όχι δίζελ αλλά με ένα μέτριο καύσιμο. Ε, δεν είναι και ο πάτος του βαρελιού που πρέπει να τον ε, τρίψεις για να βγει, είναι η μεσαία ποιότητα, ενώ άλλοι επενδύουν σε εναλλακτικά καύσιμα που βλέπουμε και με τα πρώτα ε, ε, σκάφη να κινούνται με υγροποιημένο φυσικό αέριο που είναι πολύ φιλική ε, ενέργεια και καύσιμο για το περιβάλλον και κίνητρα και προγράμματα υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενθαρρύνονται και να αυξάνουν τις επενδύσεις και να χτίζουν νέα καράβια τέτοια αεριοκίνητα για τις μεταφορές ας πούμε, πράσινη ενέργεια για τις μεταφορές. Είναι ένα πρόγραμμα που έχετε συζητήσει και εσείς. Μια άλλη τεχνολογία λοιπόν μπορεί να επιλεγεί και έχει ήδη επιλεγεί από κάποιους ε, πλειοκτήτες που είναι να καίνε μεν βαρύ καύσιμο μικρότερης ποιότητας αλλά να έχουν αυτές τις πλυντρίδες όπως είναι οι ε, καταλήτες που έχουμε στα αυτοκίνητα ε, για να ε, μειώνονται οι εκπομπές. Από αυτή τη διαδικασία την καταλητική έχουμε μικρές, περιορισμένες τοξικές ποσότητες, οι ποσότητες τοξικών καυσίμων. Δεν υπάρχει παντού σε όλα τα λιμάνια, αλλά σε κάποια λιμάνια μπορούν να αποφορτώνουν, να εκφορτώνουν αυτά τα απόβλητα, τα τοξικά, για να μην τα ε, ξεφορτώνουν στη θάλασσα. Αυτό ισχύει ήδη. Και αυτό θέλουμε να το εισαγάγουμε στη λογική της υφιστάμενης οδηγίας. Αλλά αυτό σημαίνει ότι επιβάλλουμε στους λιμένες να διαχειρίζονται ένα νέο είδος, μια νέα κατηγορία αποβλήτων που είναι πέρα από τα όσα έχουμε συζητήσει και το έχουμε συζητήσει σε βάθος και με τους ειδικούς και τους δικηγόρους μας, αλλά είναι εκτός πλέον πεδίου εφαρμογής της οδηγίας όπως προβλέπετε σήμερα αυτό και θα πρέπει λίγο να σας ζητήσουμε να κάνετε υπομονή να φέρουμε μία πρόταση που θα πρέπει να περάσει από συναπόφαση Κοινοβουλίου και Συμβουλίου έτσι ώστε να ενταχθούν και αυτές οι υποχρεώσεις με σωστό τρόπο να μπορούν τα λιμάνια να διαχειρίζονται το νέο είδος αποβλήτων. Γιατί ακόμα δεν έχει γίνει αυτό. Εμείς θα μπορούσαμε την πρόταση να την φέρουμε πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά τώρα ε, κάνουμε σε βάθος αξιολόγηση της λειτουργίας ολόκληρης της οδηγίας και όλα αυτά τα θέματα που μας απασχολούν σήμερα και αυτό ολοκληρώθηκε, αυτή η αξιολόγηση δηλαδή και κανονικά θα ε, βγει η έκθεση και θα έρθει στα χέρια σας και το Συμβούλιο και υπάρχουν και άλλα θέματα που πρέπει να ξαναδούμε ε, στην αναθεώρηση της οδηγίας. Και επειδή όλοι δεσμευόμαστε για καλύτερη νομοθεσία, το 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μελετήσει, θα, με μελέτη αντικτύπου δηλαδή τις προτάσεις που θα ε, φέρει, γιατί όλα αυτά έχουν και κόστος είτε για τους λιμένες, είτε για το περιβάλλον ή για τις ναυτιλιακές εταιρείες, ε, θα πρέπει σε βάθος να τα μελετήσουμε, οπότε και το 2017 θα έρθει πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας, η οποία θα περιλαμβάνει την επέκταση ε, των διατάξεων και σε νέα ε, είδη αποβλήτων. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ είναι που χειροκροτάμε για ε, τα όσα απαντήσατε και για τις ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επαναλαμβάνω τις ευχαριστίες. Πραγματικά ειλικρινά σε όσους μας τα παρουσίασαν. Τώρα δεν με ακούει ο κύριος Κούν όμως. Τι να κάνουμε. Αυτό έλεγα τώρα. Ευχαριστίες λέω εξ ονόματος Επιτροπής και καλό είναι να τα ακούτε κι εσείς αυτά. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ικανοποιημένοι είμαστε. Και αντιρρήσεις και ενστάσεις αν έχουμε, έχουμε προθεσμία να τις εκφράσουμε μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 27 Οκτωβρίου. Καλώς. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Εδώ πρόκειται για την παρουσίαση μιας ε, έκθεσης ε, που αφορά στο κόστος της μη ολοκλήρωσης της Ευρώπης όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών. Η Επιστημονική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μας παρουσιάσει ένα βίντεο 5 λεπτών. Αχα, das wird also später sein, höchstgrad. Όχι τώρα, θα το δείξουμε λίγο αργότερα. Ja, dann kriegt Monika Nogai das Wort für die folgende. Λοιπόν, ε, τώρα το λόγο έχει η συνάδελφός μας για την Ευρωπαϊκή Υπεραξία. Θα μας παρουσιάσει το θέμα η κυρία Μόνικα Μογκάη. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, ο κύριος Ατζόταν ε, που είναι ο ε, προϊστάμενός μου δεν μπορεί να παρίσταται σήμερα. Ε, έχει μια ε, απρόοπτη υποχρέωση. Εγώ εργάζομαι στο τμήμα Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας. Ε, η συγκεκριμένη αποστολή του τμήματος αυτού είναι να βοηθήσει τις ε, επιτροπές να ποσοτικοποιήσουν και να εντοπίσουν προτεραιότητες πολιτικών. Υποστηρίζουμε λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις αρμοδιότητες του. Υποστηρίζει, παρέχει ένα σύστημα υποστήριξης που διευκολύνει τις επιτροπές επιτροπές ε, να επεξεργαστούν ε, ε, και να καταρτήσουν εκθέσεις τη απουσία πρωτοβουλειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε τις αξιολογήσεις του τμήματός μας, σύντομα κείμενα τα οποία συνοδεύουν ε, νομοθετικού χαρακτήρα ε, εκθέσεις, ε, παρόμοιες με αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά με κατόπιν εκθέσεων πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε εκθέσεις για τομείς στρατηγικής σημασίας τους οποίους ε, υπάρχει περιθώριο περαιτέρω δράσης σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Οι εκθέσεις ε, του κόστους απουσίας της Ευρώπης προετοιμάζουν το έδαφος για μία ή περισσότερες ε, νομοθετικές πρωτοβουλίες του Κοινοβουλίου και ένας ε, τρίτος τύπος ε, προϊόντος που μπορεί να τα γνωρίζουν οι ευρωβουλευτές είναι η χαρτογράφηση, η εκθέση χαρτογράφησης του κόστους ε, της απουσίας της Ευρώπης παρουσιάζει και συγκρίνει τα διάφορα ωφέλη περαιτέρω δράσης για διάφορους τομείς ανάλογα με τις ε, αξιολογήσεις που κάνουμε, ε, με τις ε, μελέτες αξιολόγησης που σας ανέφερα και προηγουμένως. Διακόπτει ο Πρόεδρος, τρεις φορές σας είπα να κάνετε ησυχία. Αυτό που σας παρουσιάζουμε σήμερα είναι το κόστος απουσίας της Ευρώπης για την έκθεση, για την κωδικοποίηση των δικαιωμάτων των επιβατών. Θα ήθελα απλώς να σας το δείξω, κάπως έτσι είναι είναι αρκετά μακροσκελές έγγραφο. Ένα τμήμα έχει συνταχθεί εδώ ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το άλλο ε, είναι ε, αποτέλεσμα μιας μελέτης που αναθέσαμε σε έναν σύμβουλο. Ε, πρόκειται για μία έκθεση που ζητήθηκε από την Επιτροπή σας στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία με σκοπό να καθοριστεί ε, το όφελος της ύπαρξης ενός ενοποιημένου πλαισίου για τα δικαιώματα των επιβατών, ε, για το, κάτι, για το οποίο, κάτι το οποίο έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο πολλές φορές με προηγούμενες εκθέσεις του. Συγκεκριμένα η έκθεση αναλύει ε, γίνεται μια νομική ανάλυση των κενών ε, και των ασυνεπιών ε, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα, για τα δικαιώματα των επιβατών στα διάφορα, στους διάφορους τρόπους μεταφορών. Υπάρχει μια ποσοτικοποίηση των στοιχείων και κόστος που προκύπτει για τους επιβάτες και για την κοινωνία. Το κόστος αναλύεται επίσης και με ποιοτικούς όρους, αλλά η ποσοτικοποίηση είναι ε, κάτι... Ε, είναι μία από τις, ε, από, τα, από τις ιδιαιτερότητες αυτής της έκθεσης. αντί να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες στην έκθεση, κάτι το οποίο θα κάνουν οι εμπειρογνώμονές μας, θα ήθελα να σας ζητήσω να δείτε το βίντεο και το οποίο συνοψίζει τα κύρια πορίσματα της έκθεσης. Ναι, βεβαίως, λέει ο Πρόεδρος.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 Σας ευχαριστώ για το βίντεο. Θα είχα μια μικρή κριτική. Ε, νομίζω είναι κάπως υπερβολική ταχύτητα της ομιλίας. Αν το επιβραδύνατε λίγο θα ήταν καλύτερο. Sorry for Συγγνώμη, αλλά επειδή είμαι δάσκαλος εγώ το επάγγελμα, ξέρετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε. Είναι το πρώτο βίντεο που κάναμε, έτσι κινούμενα σχέδια και θα το λάβουμε υπόψη αυτό, ότι είναι γρήγορα μιλή. Αν μου επιτρέπετε να δώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονες τώρα για να σας τα αναλύσουν περισσότερο, για το, ε, ποια είναι τα ευρήματα της ένας. Και πάλι σας επιτρέπω. Good afternoon. So my name is Natalie Καλησπέρα, Ναταλή Μορένς. Ε, με τη συνάδελφό μου την Ανιέσκα Μαρκόφσκα θα παρουσιάσουμε με λίγο περισσότερες ε, λεπτομέρειες, ε, λίγο, περισσότερο, λίγο περισσότερα από αυτά που είδατε στο βίντεο. Ελπίζω να σας χρησιμεύσουν αυτά που θα ακούσετε. Θα συζητήσουμε λοιπόν ε, το πλαίσιο των δικαιωμάτων των επιβατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως ε, τα κενά που βλέπουμε στην ε, ενωσιακή νομοθεσία και μετά η συνάδελφός μου θα σας μιλήσει για τη μεθοδολογία που ακολουθήσαμε για την αξιολόγηση του κόστους αυτών των κενών. Ε, και να μπορούμε, να μπορούμε μετά να προχωρήσουμε και, για, και στο είδο της κωδικοποίηση που προτείνουμε. Όπως γνωρίζετε, είναι βασικό τομέα οι μεταφορές για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά πολλούς ε, επιβάτες ετησίω. 800 ε, εκατομμύρια επιβάτες ε, με χερσαία μέσα μεταφορά στο χρόνο και 400 εκατομμύρια διαθαλάσσεις ε, πρέπει να κωδικοποιήσουμε τα δικαιώματά τους με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι λιγότερα τα προβλήματα που θα αντιμετωπίζουν και τα εμπόδια που θα βρίσκουν στο δρόμο τους. Υπάρχουν, υπάρχει νομοθεσία σε διάφορες χρονικές στιγμές ανάλογα ανάλογα με το είδος της μεταφοράς και υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα προστασίας ε, σε αεροπορικές ε, ε, μεταφορές, σε μεταφορές ε, ε, με το σιδηροδρομικές μεταφορές και επομένως υπάρχουν πάρα πολλά κενά. Να σας δώσω μια γενική θεώρηση καταρχάς των 10 βασικών ε, δικαιωμάτων που υπάρχουν και των κενών που έχουμε εντοπίσει. Θα ήθελα καταρχάς να σας πω τι εννοούμε κενό. Κενό εννοούμε ότι η νομική διάταξη δεν ορίζεται σε κάποιο τομέα, στους, σε διάφορους τρόπους μεταφορές ή στην πράξη σημαίνει ότι με έρευνα ανακαλύψαμε ότι τα δικαιώματα δεν ε, εφαρμόζονται στην πράξη. Και τι λέμε ασυνέπεια. Λέμε ότι υπάρχει διαφορετικό επίπεδο προστασίας ε, για, έναν, ε, για, τους, για τους επιβάτες ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς. Για παράδειγμα, ε, ε, στη νομοθεσία για τις αεροπορικές μεταφορές δεν αναφέρεται τίποτε όσον αφορά την εξασφάλιση της, ε, της τοποθέτησης του επιβάτη σε ένα νέο δρομολόγιο αν υπάρξει για κάποιο λόγο κάποια κύρωση. Κάτι το οποίο δεν ισχύει για τα σιδηροδρομικά. Είναι, διαφορετικά, λοιπόν, είναι διαφορετικό το επίπεδο των δικαιωμάτων και το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των ατόμων με ε, μειωμένη κινητικότητα. 84 κενά και ασυνέπειες έχουμε εντοπίσει στην υφιστάμενη νοσιακή νομοθεσία και αυτά τα κενά και οι ε, συνέπειες έχουν να κάνουν με το δικαίωμα πληροφόρησης, το δικαίωμα ε, υποστήριξης και μάλιστα το δικαίωμα που παραβιάζεται περισσότερο είναι αυτό της πληροφόρησης το δικαίωμα στην αποζημίωση ε, το δικαίωμα δηλαδή του ε, επιβάτη να γνωρίζει τα δικαιώματά του είτε για την τιμολόγηση είτε για το ε, δικαίωμα υποστήριξης και αποζημίωσης. Είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό των επιβατών που υποβάλλουν καταγγελία ή ζητούν αυτά τα οποία δικαιούνται. Επομένως είναι, ένα, είναι προβληματική, προβληματικό αυτό το δικαίωμα συγκεκριμένα και πρέπει πραγματικά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να ενισχύσουμε. Να περάσουμε τώρα στο κόστος των κενών αυτών. Θα σας μιλήσει η συνάδελφος γι' αυτά. Όσον αφορά τη μεθοδολογία αξιολόγησης του κόστους, ε, επειδή είχαμε περιορισμό ε, στη μεθοδολογία και στα ε, είχαμε περιορισμό στα δεδομένα που είχαμε στη διάθεσή μας, δεν κατέστη εφικτό να υπολογίσουμε όλα τα στοιχεία του κόστους σε σε νομισματικούς ε, όρους ε, και όπως βλέπετε στον πίνακα, αυτά, αυτοί είναι οι τέσσερι τομείς ε, που μπορέσαμε να ποσοτικοποιήσουμε. Η διαφάνεια, η ποιότητα της υπηρεσίας, ε, η επιβολή και η διατροπικότητα, στους οποίους τομείς καταφέραμε να κάνουμε μία αξιολόγηση σε νομισματικούς όρους. Και οι έξι τομείς ε, έχουν αναφερθεί στην έκθεση Μπαχ ε, και έχουν ε, υπάρξει αντικείμενο ποιοτική αξιολόγηση και όταν λέω ποιοτική εννοώ και η ιεράρχηση των συνεπειών και κατηγοριοποίησή του αναλόγως με το αν η συνέπεια ήταν σοβαρή, λιγότερο σοβαρή ή όχι σοβαρή. Όσον αφορά τώρα το κόστος, βασιζόμαστε σε, ε, στη γενική έννοια του ε, καθαρού κοινωνικού κόστους, ε, δηλαδή μεταφορές μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων φορέων δεν ελήφθησαν υπόψη ως κοινωνικό κόστος. Και μιλάω τώρα για το ποσό της αποζημίωσης, για παράδειγμα, που από τη μία αποτελούν ένα όφελος για τους επιβάτες, από την άλλη όμως είναι ένα κόστος, ένα επιπλέον κόστος για ε, τους ε, μεταφορείς. Αυτό λοιπόν δεν συμπεριλαμβάνεται στην ε, εκτίμηση. Τώρα, πώς έγινε υπολογισμό του κόστους, δεν θα σας πω λεπτομέρειες γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Να σας δώσω όμως ένα παράδειγμα. Μία σημαντική κατηγορία ήταν ο χρόνος που χάνεται λόγω της έλλειψης διαφάνειας. Επί και εμπροκειμένου ασχοληθήκαμε με τον ε, τομέα των ε, εναερίων μεταφορών, όπου πολύ συχνά ε, διαπιστώνουμε ότι οι επιβάτες δεν έχουν σαφή διαφανή πληροφόρηση από την αρχή της διαδικασίας κράτησης σε σχέση με την τιμή και το είδος των υπηρεσιών που συμπεριλαμβάνει η τιμή της υπηρεσίας που να τους επιτρέπει να συγκρίνουν την τιμή αυτή με άλλες προσφορές. Οι επιβάτες λοιπόν απλώς χάνουν χρόνο που θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν για, με πολύ πιο παραγωγικό τρόπο. Ε, κάναμε λοιπόν μια εκτίμηση της αξίας του χρόνου που χάνεται, ε, πολλαπλασιάζοντας την εκτίμηση του αριθμού των ωρών ε, που χάνονται, σε αυτές τις περιπτώσεις επί μιας συγκεκριμένης τιμής ανά Επίσης, εκτιμήσαμε το νομισματικό κόστος στην περίπτωση της έλλειψης υποστήριξης. Έχουμε κάνει και την αντίστοιχη εκτίμηση στον τομέα της ε, επιβολής ο χρόνος που χάνεται κατά τη διάρκεια της, του, ε, της διαχείρισης μιας καταγγελίας, αυτές οι διαδικασίες είναι πάρα πολύ ε, μακροχρόνιες γιατί δεν υπάρχουν επαρκείς και διαφανείς πληροφορίες και επίσης κάναμε και την εκτίμηση του κόστου χρόνου, του κόστος χρόνου ε, λόγω της ε, απώλειας χρόνου όταν αλλάζει κανείς τρόπο μεταφοράς, λόγω της διατροπικότητας δηλαδή αυτό μπορεί να θεωρείται ελάχιστη, ένα ελάχιστο, μια ελάχιστη εκτίμηση και αυτό ισχύει γιατί δεν μπορέσαμε να συνυπολογίσουμε όλους τους τομείς, όλα τα στοιχεία του κόστους σε όλους τους τομείς και μιλάω ειδικότερα για τον τομέα των οδικών μεταφορών και των ε, ε, θαλασσίων μεταφορών ή των, μεταφορών σε πλωτές οδούς, ε, γιατί τα δεδομένα απλώς δεν ήταν διαθέσιμα. Τα περισσότερα δεδομένα που είχαμε στη διάδοση μας αφορούσαν ε, τις εναέριες μεταφορές. Όπως ε, είδατε, το συνολικό κόστος της απουσίας της Ευρώπης κατ' έτος έχει εκτιμηθεί στα 355 εκατομμύρια ευρώ ετησίως το υψηλότερο κόστος ε, στο τομέα, στον τομέα της διατροπικότητας και της ε, διαφάνειας. Επομένως, αυτό το κόστος αυτούς τους δύο τομείς είναι άνω των 100 εκατομμυρίων ε, ευρώ κατ' έτος, ενώ στον τομέα της επιβολής έχουμε εκτιμήσει το κόστος στα περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ κατ' έτος και στην ε, ποιότητα της υπηρεσίας ε, η εκτίμησή μας ανέρχεται σε 20 εκατομμύρια ευρώ κατ' έτος περίπου. Δεν σημαίνει ότι το κόστος μπορεί πάντοτε να εκφράζεται κατά αυτόν τον τρόπο. Ε, ε γι' αυτό έχουμε και μία πολύ εκτενή ποσοτική ανάλυση Για παράδειγμα υπάρχει και το, το ψυχολογικό ε, στοιχείο, το άγχος, ε, που είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο να το εκφράσουμε σε όρους κόστους. Ε, υπάρχουν βέβαια κάποιες, θε, τι, κάποιες θεμελιώδεις τιμές που έχουν να κάνουν για παράδειγμα με την διάκριση ή την υποστήριξη ατόμων μειωμένης κινητικότητας και υπάρχει επίσης και μεγάλο φάσμα ε, άλλων ε, οικονομικών παραμέτρων όπως είναι ο ανταγωνισμός, ε, ο αντίκτυπος στο περιβάλλον, η απώλεια χρόνου και η αναποτελεσματικότητα που προκύπτει από αυτό δεδομένου ότι ο χρόνος αυτός θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιηθεί παραγωγικότερα από τους χρήστε. Επίση, διαπιστώνουμε ότι κάποιοι από τους επιβάτες ε, που έχουν απογοητευτεί ε, από τις δημόσιες μεταφορές ε, θα χρησιμοποιήσουν τελικά το αυτοκίνητό τους αντί για τα μέσα μεταφορά στα δημόσια. now we, we look over... Πέντε τώρα επιλογές κωδικοποίησης, ε, κάτι το οποίο προτείνουμε στην έκθεσή μας. Ε, τι εννοούμε κωδικοποίηση. Είναι ένας ε, τεχνικός όρος του να τα συμπεριβάλλουμε όλα αυτά σε μία πράξη, όλη η νομοθεσία που υπάρχει να συμπεριληφθεί σε μία πράξη χωρίς ουσιαστικές αλλαγές. Αυτό είναι η πρώτη επιλογή ουσιαστικά θα σήμαινε ότι όλη η νομοθεσία θα συμπεριληφθεί σε μία πράξη χωρίς τροποποίηση όμως ε, δεν θα ε, έχει ως αποτέλεσμα ιδιαίτερη εναρμόνιση, όμως θα διευκολύνει την ε, πληροφόρηση και τη διαφάνεια της πληροφόρησης. Μία καλύτερη επιλογή θα ήταν ενδεχομένως η τροποποίηση της νομοθεσίας πριν περάσουμε στην κωδικοποίηση, οπότε κάθε νομοθεσία θα αναθεωρηθεί για να καλυφθούν αυτά τα κενά που αναφέραμε. Αυτή είναι μια διαδικασία βέβαια που θα είναι πολύ μακροχρόνια και είναι βέβαια και υψηλό το κόστος εφαρμογής αυτής της εναλλακτική επιλογής ε, και αν ήταν χαμηλό το κόστος μπορεί να μην καλύψει τότε κάποια κενά. Τρίτη επιλογή είναι βελτιωμένη και πιο αποτελεσματική κωδικοποίηση που είναι η αναδιατύπωση βεβαίως, κάτι το οποίο στην ουσία σημαίνει ότι ενώ θα έχουμε μία πράξη ενιαία, πρέπει να γίνει και η διαδικασία της ε, αναθεώρησής τους κατά τη διάρκεια της κωδικοποίησης. Οπότε αυτό πρέπει να γίνει με το υψηλότερο επίπεδο εναρμόνισης για να έχει νόημα και να καλύψει έτσι τα ε, περισσότερα κενά. Χρειάζεται βέβαια μεγάλη προσπάθεια για να γίνει κάτι τέτοιο, μια τέτοιου είδους, ένα τέτοιο εγχείρημα να ε, διατύπωσης. Και βέβαια το κόστος εφαρμογής θα είναι υψηλό για τα κράτη-μέλη. Μία ακόμη επιλογή είναι το κοινό πλαίσιο αναφοράς, που είναι ουσιαστικά ένα πακέτο εργαλείων που θα διευκρινίσουν κάποιους όρους, κάποιους ορισμούς, κάποιες έννοιες ε, και ε, αυτό ε, βέβαια χάρη διαφάνειας και σαφήνειας στην νομοθεσία δεν θα έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο βέβαια, ε, ούτε θα προκύψουν νέα ε, δικαιώματα, όμως τουλάχιστον αν υπάρχει αυτό το κοινό πλαίσιο αναφοράς μπορεί να συνδυαστεί με τη δεύτερη εναλλακτική επιλογή και η τελευταία επιλογή είναι μία χάρτα ε, που θα μπορούσε ως αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ γνωστά τα δικαιώματα των επιβατών. Είναι ε, πολύ πιο εύκολη έτσι η γνωστοποίηση των δικαιωμάτων αυτών. Βέβαια είναι μη δεσμευτικό αυτό το μέσο και δεν θα ε, διευκολύνει ε, αναθεώρηση της νομοθεσίας. Μπορούμε βέβαια να συνδυάσουμε τις διάφορες επιλογές, για παράδειγμα αναδιατύπωση και χάρτα. Αυτό θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη εναρμόνιση και καλύτερα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ να απαντήσω σε ερωτήσεις. Λοιπόν, καταρχήν ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ομιλίες και για το βίντεο. Τώρα παρακαλώ αν θέλετε μπορείτε να ε, κάνετε ερωτήσεις. Ο κύριος Γκόλνης. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και το βίντεο και εξηγήσεις που ακούσαμε, πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ε, όμως εγώ προβληματίζομαι λίγο για το τελικό αποτέλεσμα. Διότι εξ όσων κατάλαβα, τα δεδομένα για το κόστος της μη Ευρώπης δεν ε, λαμβάνουν υπόψη την αύξηση του κόστους για ε, τις εταιρείες που τα διαχειρίζονται ε, όλα αυτά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και κάπως ε, έτσι προσβάλλεται η αξιοπιστία της ε, έρευνας και της μελέτης. Τι εννοώ, η καλύτερη προσβασιμότητα ας πούμε στο τρένο για τους ε, ανθρώπους με αναπηρίες έχει ένα κόστος το οποίο είναι θεμητότατο και το οποίο θα πρέπει η κοινωνία να επομίζεται και οι μεταφορικές εταιρείες, εταιρείε, δηλαδή στο όνομα της αλληλεγγύης, της εις πρόσβαση όλων των ε, επιβατών, αρτιμελών ή αναπήρων. Αλλά εγώ προβληματίζομαι ε, ε, ως προς τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η έρευνα. Έχετε υπολογίσει το κόστος αυτό για τις διάφορες εταιρείες συγκοινωνιών. Ο Πρόεδρος. Το κόστος για τα άτομα με αναπηρία. Το αναλαμβάνουν εκείνοι που δεν είναι ανάπηροι. Και εγώ σας λέω ότι εγώ με χαρά πληρώνω γιατί χαίρομαι κάθε μέρα που δεν έχω αναπηρία. Ναι, υπάρχουν όμως κάποιες δρομικές ή αεροπορικές εταιρείες που λέγουν «Εμένα δεν με ενδιαφέρει, εγώ θέλω να έχω φτηνά εισιτήρια και θέλω και πλεονεκτήματα και αν είναι μερικοί ε, ε, ε, με αναπηρία δεν τους παίρνουμε». αυτό είναι τρομακτικό γιατί όλη η κοινωνία πληρώνει και οι άλλοι βγάζουν κέρδη. Είναι απαράδεκτο. Αυτό χρειάζονται δίκαιοι και ίσοι κανόνες για όλους. Ένα δεύτερο σημαντικό. Στις σιδεροδρομικές μεταφορές. Βεβαίω θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης όλοι οι άνθρωποι με αναπηρία, οι πάντες όμως να ισχύει για όλους αυτό και δεν θα πρέπει κανένας να ξεφεύγει από τις ευθύνες του. Και καλό είναι να έχουμε αυτή την ανάλυση. Ενώ στα αεροπλάνα δεν έχουμε ε, κανένα, ε, καμία υπηρεσία που να μπορεί κανείς να προσφεύγει για την επίλυση διαφορών. Στη Γερμανία υπάρχει αυτό στο σιδηρόδρομο 85% μπορείς να πας. Υπάρχει ε, ένας διαμεσολαβητής και δεν υπάρχουν ουσιαστικά διενέξεις. Και έχει αναλυθεί ότι μόνο το 1% εκείνων που δικαιούνται ε, αποζημίωση δηλαδή ε, ε, στις αεροπορικές μεταφορές όταν έχουν καθυστερήσεις αεροπλάνα κτλ. Δεν το κάνουν. Εγώ ξέρω μια γερμανική αεροπορική εταιρεία που δεν κάνει τίποτα. Και στις λίγες περιπτώσεις το 1% που προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, λίγο πριν εκδοθεί η δικαστική απόφαση λένε Ωραία, το δεχόμαστε γιατί δεν θέλουν να έχουν δικαστική απόφαση, καταδικαστική ουσιαστικά. Αυτή η πρακτική είναι τελείως αντικοινωνική και δεν επιτρέπεται εμείς να το δεχτούμε. 355 εκατομμύρια ποιος θα πληρώνει αυτά. Η κοινωνία, οι άλλοι επιβάτες και όποιο θέλει να κερδοσκοπεί είναι αυτές οι εταιρείε, οι αεροπορικές ή οτιδήποτε, οι οποίες δεν επιτρέπεται να επιδεικνύουν τέτοια συμπεριφορά. Είναι απαράδεκτη. Ήθελα να τα πω αυτά. Κάτι λέει ο κύριος Βαντεκάμπ. Και με μικρόφωνο τώρα. Περίμενα μια στιγμή να ζητήσει λεφτά το ότι θα και δίσκο δηλαδή, όπως στην εκκλησία, να κάνεις έρανο. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ε, κύριε Κράμερ. Αυτό δεν ήταν ε, ο στόχος της μας. δηλαδή να ερευνήσουμε το κόστος για τα σκάφη που προσφέρουν βοήθεια, ή πληροφορίες, ή ε, το επίπεδο διαφάνειας ε, το οποίο είναι αναμενόμενο στη σύγχρονη κοινωνία. Είδαμε λοιπόν ότι μόνο το 17% των ε, των εταιριών δίνουν πληροφορίες με τρόπο διαφανή. Ε, άρα δηλαδή το θέμα είναι ότι θα πρέπει να δούμε, να υπολογίσουμε το κόστος ε, για να προσφέρονται υπηρεσίες σε ένα επίπεδο ποιότητας το οποίο είναι το αναμενόμενο στην κοινωνία μας. Είναι λοιπόν αλήθεια ότι μια τέτοιου είδους ε, ανάλυση μπορεί να είναι συμπληρωματική, αλλά αυτό δεν είναι το, ο βασικός στόχος ε, της αναλυσής μας. Εμείς έχουμε εστιάσει την προσοχή μας ε, στο κοινωνικό κόστος της μη Ευρώπης ε, και επίσης διαπιστώσαμε το κόστος αυτό υπολείπεται κατά πολύ του αναμενόμενου και του βέλτιστου. Πολύ ωραία λέει ο Πρόεδρος. Τότε παρακαλώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοποθετηθεί ο κύριος Κόλσον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα αυτό που θέλω να πω ευθύς εξ αρχής είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι δεσμευμένη να διασφαλίζει, να προστατεύει και να αναπτύσσει τα δικαιώματα των επιβατών. Και η μελέτη προσφέρει μια πολύ καλή γενική εικόνα των κενών που υπάρχουν των ασυνεπιών ε, στις, στο, στις νομοθεσίες ε, για τα δικαιώματα των επιβατών για όλα τα μέσα μεταφοράς. Βεβαίως, με κάθε σεβασμό στους ε, συντάκτες της ε, μελέτης, εμείς θεωρούμε ότι μια μελέτη για την δυνατότητα εφαρμογής και τις επιπτώσεις της μελέτης αυτής θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις διατάξεις και τις αρχές που διέπουν τα δικαιώματα των καταναλωτών με στόχο την εναρμόνιση των δικαιωμάτων ε, σε όλα τα μέσα μεταφοράς. Ε, θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω με κάποια γενικής φύσεως σχόλια. Υπάρχουν λοιπόν ασυνέπειες όπως σας είπα και κενά τα οποία αποδυναμώνουν την ποιότητα της έκθεσης. Παραδείγματο χάρη διαπιστώσαμε μία σειρά λατών που αφορούν στην περιγραφή των ε, ρόλων ε, που έχουν σχέση με την εφαρμογή της ε, νομοθεσίας. Παραδείγματο χάρη τα παραδείγματα της ανωτέρας βίας δεν ευστατούν ή το δικαίωμα σε αυτό αφορά και τις μεγάλες καθυστερήσεις και δεν αναφέρεται, αναφέρεται το αντίθετο. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για να υπολογιστεί το κόστος από το ότι δεν υπάρχει ένα ενοποιημένο πλαίσιο για τα δικαιώματα των επιβατών, αυτό δεν είναι σαφές. Οι παραδοχές πίσω από τους υπολογισμούς δεν είναι πιστικές και μάλιστα δεν σχετίζονται και με τα δικαιώματα των πολιτών στο τρέχον νομοθετικό πλαίσιο. Παραδείγματο χάρη το κόστος των 130 εκατομμυρίων ευρώ που οφείλεται στην έλλειψη διατροπικότητας είναι παραπλανητικό ε, γιατί ανάγεται περισσότερο ε, στο ότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σύστημα ticketing. Αυτό όμως δεν μπορεί να επιληθεί με απλή κωδικοποίηση της νομοθεσίας περί δικαιωμάτων επιβατών. Πάντως, ε, κατά την άποψή μας, η μελέτη τελικά δεν κατορθώνει να καταδείξει ότι η κωδικοποίηση όλων των νομοθετημάτων για τη δικαιώματα των πελατών πελατών είναι η μόνη εφικτή λύση για να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και συμφωνούμε ότι υπάρχουν αδυναμίες ως προς τα δικαιώματα των επιβατών και υπάρχουν δύο βασικά θέματα που ε, ελέγχονται στην έκθεση κενά, ασυνέπειε στην κείμενη νομοθεσία για τα δικαιώματα των επιβατών και έλλειψη νομοθετικού πλαισίου που να αφορά στα διατροπικά ταξίδια. Για το πρώτο, η μελέτη δεν προσφέρει σαφή στοιχεία για να αποδείξει το γιατί η κωδικοποίηση είναι η πιο ε, κατάλληλη λύση για να ε, καλυφθούν τα κενά που έχουν εντοπιστεί στην νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα, η κωδικοποίηση δεν είναι απαραίτητα η καλύτερη επιλογή και μάλιστα δεν είναι και εφικτό να ε, καλυφθούν κάποια κενά ακόμα και αν έχουν εντοπιστεί. Το γεγονός ότι κάποια κενά αφορούν όλα τα μέσα μεταφοράς, αυτό από μόνο του δεν αιτιολογεί την κωδικοποίηση ή την αναπομπή. Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσα, ξεχωριστά μέσα από τροπολογίες. Η ύπαρξη λοιπόν διαφορετικών κανόνων μπορεί να δικαιολογηθεί με αντικειμενικές διαφορές ε, όσον αφορά στα μέσα μεταφοράς και επίσης και από το γεγονός ότι ορισμένοι κανόνες που κυρίως ε, έχουν σχέση με την αστική ευθύνη αυτά προέρχονται από εθνικές συμβάσεις που δεν μπορούν να τροποποιηθούν. Άλλα προβλήματα ανάγονται στην ίδια η νομοθεσία και στο ότι δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία αυτή. Αυτό είναι διαφορετικό αλλά δεν λύνεται με την κωδικοποίηση. Όσον αφορά στην έλλειψη νομοθετικού πλαισίου για τα ε, διατροπικά ε, ταξίδια γνωρίζουμε πολύ καλά το ότι θα ήταν χρήσιμο να υπάρχουν κανόνες για να προστατεύονται οι επιβάτες οποτεδήποτε κάνουν ε, τέτοιου είδους ταξίδια ή έστω και με ένα μέσο μεταφοράς. Ωστόσο, η τροποποίηση όλη τη κείμενη νομοθεσίας θα ε, ε, ενήχε τον κίνδυνο να ξανανοίξουν μακροσκελείς συζητήσεις και διαπραγματεύσεις και ενδεχομένως αυτό ε, θα σήμαινε αποδυνάμωση όλου του κοινωτικού κεκτημένου. Το βλέπουμε ήδη ε, για το πώς, βλέπουμε πώς συζητάει το Συμβούλιο τα θέματα των δικαιωμάτων των επιβατών. Για το λόγο αυτό μάλλον ε, είμαστε υπέρ άλλων ε, λύσεων όπως νέα νομοθεσία για τα δικαιώματα των επιβατών στις διατροπικές μεταφορές. Τέλος θα έλεγα ότι ο ίδιος στόχος, η βελτίωση δηλαδή της προστασίας των επιβατών ε, θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς να διακυβευτεί το σύνολο του κοινοτικού κεκτημένου μέσω άλλων δραστηριοτήτων. Όπως είναι ε, να πληρωθούν τα υφιστάμενα νομικά κενά που έχουν να κάνουν με τη διατροπικότητα με διαφορετική ξεχωριστή νομοθετική πρωτοβουλία και ε, όταν αναθεωρηθεί η κείμενη νομοθεσία να συμπεριλαμβάνεται όταν είναι αυτό δυνατό μια ειδική διάταξη ή ειδικέ διατάξεις ώστε να εξασφαλίζονται ίσοι κανόνες παιχνιδιού και να φορούν όλα τα μέσα μεταφοράς και μέσω της ε, σωστής υλοποίησης σιγά σιγά να συγκλίνει η νομοθεσία. Είναι περίπλοκα αυτά τα θέματα και δεν έχουν και σαφήνεια πολλές φορές οι νομοθετικές διατάξεις. Αυτό λύνεται με ε, ερμηνευτικές ε, κατευθυντήριες γραμμές όπως έγινε για ε, επιβάτες με περιορισμένη κινητικότητα ή για επιβάτες σιδηροδρόμων πρόσφατα. Αλλά με την οδηγία αυτή θα πρέπει να επιμείνουμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις τους και να ε, προωθούν και να εφαρμόζουν και να επιβάλλουν τα δικαιώματα των επιβατών σε εθνικό επίπεδο. Συμφωνούμε ότι υπάρχουν αδυναμίες και με τη διαπίστωση, αλλά διαφωνούμε με τον τρόπο που προτείνεται με ΑΙ να επιληθούν αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ μετά από αυτή τη διάλεξη θα πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στις δύο συγκήτρες να απαντήσουν σε όλα αυτά που είπατε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. I just have to clarify. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι εμάς μας ζήτησαν να δούμε πώς μπορεί να γίνει η κωδικοποίηση. Συμφωνώ ότι μπορούν να υπάρχουν και άλλες δυνατότητες, αλλά οι επιλογές ε, κωδικοποίησης ε, περιλαμβάνουν και ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς που μπορεί να θεωρηθεί και κατευθυντήρια γραμμή Βεβαίω υπάρχουν και άλλοι τρόποι να βελτιωθεί η εφαρμογή όλων αυτών και η νομοθεσία. Αλλά εμάς μα ζήτησαν να πούμε για την κωδικοποίηση. Λάβαμε βεβαίω υπόψη ε, τη διαφορά ε, ανάμεσα στα διάφορα μέσα μεταφοράς και όταν υπάρχουν αντικειμενικές ε, διαφορές δεν τις θεωρήσαμε ούτε ελλείψεις, ούτε κενά, ούτε ασυνέπειες. Αν έχετε άλλο σχόλιο για κάποιο λάθος που κάναμε, παρακαλώ να μας ενημερώσετε και θα το διορθώσουμε. Επίσης, πολλά από αυτά που είπατε και τα προβλήματα που έχουν ανακύψει έχουν να κάνουν με την εφαρμογή και την υλοποίηση. Δεν απαντώνται από την κωδικοποίηση, αλλά θα μπορούσε να βοηθήσει η κωδικοποίηση για να ενισχυθεί η εθνική υλοποίηση. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Εμείς ήμασταν περιορισμένοι στη μελέτη μας γιατί μας ζητήθηκε να μελετήσουμε, επαναλαμβάνω, την κωδικοποίηση. Και ελπίζω να σας κάλυψα με την απάντησή μου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βαντεκάμπ. Πρόεδρε, πολύ ενδιαφέρον το απόγευμα. Ε, πολύ ωραίες συζητήσεις κάνουμε. Θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για ένα έγγραφο της δικής μας υπηρεσίας. Ε, έτσι, αυτό, αυτή η έκθεση που μας παρουσιάστηκε είναι δική μας και την έχουμε αναθέσει εμείς. Θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας στείλει γραπτό σε αυτό το σχόλιο που διάβασε εδώ. Και να πω το εξή ακόμα. Είναι πολύ ωραίο και ε, είναι να λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν χρειάζεται κωδικοποίηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το λέει αυτό, άκουσον άκουσον. Και ε, βέβαια δεν μπορούμε τώρα να συμφωνήσουμε, αλλά ε, οι δύο κυρίες έκαναν την έρευνα αυτή και είναι δική μας υπηρεσία και υπάρχει και η μελέτη σκοπιμότητας. Έχουν σύνδεση αυτά τα δύο. Ε, φαίνεται να είναι το ίδιο, αλλά δεν είναι. Το ένα είναι εκ των προτέρων, το άλλο είναι εκ των υστέρων. Αυτό στο μέλλον τι σχέση θα έχει μεταξύ του. Χρειάζεται λίγη προσοχή. Να μην τα κάνουμε όλα διπλά, να τα ψάχνουμε. Δηλαδή να κάνουμε μία έκθεση και μελέτη αντικτύπου και μετά αξιολόγηση. Δεν θέλουμε να κάνουμε διπλό έλεγχο. Α, ο κύριος Κόχ. Δεν σας είδα. kein problem, wenn ich... Ε, εντάξει, δεν είναι πρόβλημα. Ήμουνα στην άκρη και δεν με είδατε. εγώ έχω μία ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ως εισηγητής ε, για το ticketing, το διατροπικό, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε, αλλά έχετε συγκεκριμένες απόψεις, ε, έτσι ένα χρονικό ορίζοντα ε, για το πότε θα υποβληθούν συγκεκριμένες προτάσεις, γιατί αυτό το έχουμε ζητήσει στην έκθεσή μου. Έχουν τεθεί λοιπόν ερωτήματα, δεν θέλουμε να κάνουμε διπλές έρευνες όταν αυτό είναι περιττό, αλλά αν καταλήγουμε σε διαφορετικά συμπεράσματα, είναι καλό να υπάρχουν δύο εκθέσεις και εμείς καλούμεθα να αποφασίσουμε ποιος έχει έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο και γι' αυτό λοιπόν σήμερα το απόγευμα είχαμε μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Επιτροπή ε, να τη ρωτήσω κατά πόσον αυτά που μας είπατε μπορείτε να μας τα δώσετε και σε γραπτή μορφή γιατί τα θέλει οπωσδήποτε ο κύριος Βαντεκάμπ αλλά ε, εντάξει αν θέλετε μπορείτε να τοποθετηθείτε από αυτού. Ναι, βεβαίως. Τα σχόλια αυτά μπορούν να σας αποσταλούν γραπτό, βεβαίω. Ευχαριστώ. Και για το ενίο εισιτήριο, δεν ξέρω εσεί ποιο θα μας τα πει τώρα, ποιος θα απαντήσει σε αυτό. Αν έχετε συγκεκριμένα σχέδια ήδη, γραπτό και αυτό. On travaille actuellement, on commence à... Ε, αυτό τον καιρό ακριβώς επεξεργαζόμαστε ε, μία νομοθετική πρόταση για τη διατροπικότητα. Εγώ ε, πάντα δυσκολεύομαι να σας δώσω χρονοδιάγραμμα γιατί το, με το Better Regulation και όλα αυτά παίρνουν χρόνο οι διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος θα ήταν όμως τέλη του 2017 να μπορούμε να κάνουμε αυτή την πρόταση. Και γιατί νωρίτερα θα ρωτήσω, πράγμα που ρώτησα και προηγουμένως. Συμφωνούμε να απευθύνουμε μια έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μήπως να επιτάχυνε κάπως. Καλώ. Dann, äh, λοιπόν αυτό το θέμα. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρουσιάσεις, για το φιλμάκι που είδαμε, το βίντεο και όλα αυτά τα ωραία που μας είπατε. Και πάμε στο επόμενο θέμα, ε, που είναι η έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα εξαιρέσει χορηγούμενε από τα κράτη-μέλη δυνάμει του κανονισμού 1371 του 2007 σχετικά με τα δικαιώματα και τι υποχρεώσει των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών. Τότε ήταν ο Ντέρκ Στέρξ, θυμάστε, εισηγητή πριν από 8 χρόνια, το είπα και το πρωί, αλλά εδώ ε, ε, θέλουμε να ακούσουμε ε, με μεγάλο ενδιαφέρον πώς εξελίχθηκε η κατάσταση. Θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Ζαν Κολσόν, και μετά στα μέλη της Επιτροπής μας. Yes, thank you very much, Mr. Chairman. I will, uh, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγγλικά θα τα πω ε, σύντομα για την έκθεση. Ε, και από τότε που εκδόθηκε η έκθεση αυτή... Όπως γνωρίζετε, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εξαιρέσεις ε, για κάποιους σιδηροδρόμους, έχουν εξαιρέσεις για εσωτερικές γραμμές ε, μεγάλης ε, απόστασης μέχρι το 2024 για σιδηροδρομικές υπηρεσίες. Μπορούν να το κάνουν για αστικό, περιαστικό και περιφερειακό σιδηρόδρομο για μια περίοδο αόριστη και επίσης για συγκεκριμένα δρομολόγια που ε, εκτελούνται εκτός ε, επικράτειας Ευρωπαϊκής Ένωσης και πάλι χωρίς χρονικό ε, περιορισμό. Εμείς κάναμε την έκθεσή μας αυτή στις 3 Δεκεμβρίου του 2009, πριν από 6 χρόνια σχεδόν. Ποια ήταν η κατάσταση λοιπόν στις 3 του 9 και ποια είναι στις 3 του 15 μόνο τέσσερα κράτη-μέλη, τέσσερα, εφαρμόζουν πλήρως τον κανονισμό. Δανία, Ιταλία, κάτω χώρες, Σλοβενία. 22 κράτη-μέλη έχουν εξαιρέσεις ε, σε επικυλωμενο βαθμο βαθμό. Πέντε κράτη-μέλη, για παράδειγμα, είχαν πλήρεις εξαιρέσεις και εφαρμόζουν μόνο τα, τις δεσμευτικές. Η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Λετωνία και η Ρουμανία. Οπότε μόλις το 36% όλων των υπηρεσιών ε, σε ό,τι αφορά επιβάτη ανά χιλιόμετρο είχαν μηδενικές εξαιρέσεις. Θα μπορούσα και πάλι να αναφέρω όλα τα κράτη-μέλη που έχουν όλες αυτές τις εξαιρέσεις Αυτό που είναι σαφές από την έκθεση είναι ότι έχουμε μία κουρελού ε, διαφορετικών κανόνων που σημαίνει ότι ε, τα κράτη-μέλη ε, δεν επιτρέπουν στους επιβάτες να κάνουν χρήση των δικαιωμάτων τους, δεν υπάρχουν ίσοι κανόνες για το σιδηρόδρομο, δεν υπάρχει διαφάνεια στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα που δημιουργεί ε, ε, ε, που είναι στρέβλος του ανταγωνισμού στο κάτω-κάτω. Τι αλλαγές έχουν γίνει. Δεν είναι και πάρα πολλέ από τις 3 Δεκεμβρίου 2014, πέντε χρόνια μετά. Μόνο πέντε κράτη-μέλη τώρα εφαρμόζουν τον κανονισμό χωρίς καμία εξαίρεση. Εκτός από τα τέσσερα που ανέφερα προηγουμένως, ήρθε να προσθεθεί και το Βέλγιο. Πέντε κράτη-μέλη λοιπόν πλέον εφαρμόζουν απολύτως και πλήρως τον κανονισμό. Η δε Γαλλία ε, αφαίρεσε τις εξαιρέσεις για εγχώριες υπηρεσίες μεγάλων αποστάσεων. Δηλαδή εφαρμόζει τον κανονισμό όχι μόνο για τις διεθνείς υπηρεσίες αλλά και για τις εγχώριες μεγάλων αποστάσεων, επαναλαμβάνω. Εκτός από αυτές τις δύο αλλαγέ, ε, το Βέλιο και τη Γαλλία λοιπόν, και ενδεχομένω το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί το σκέφτεται, μήπω εφαρμόσει τον ε, κανονισμό ευρύτερα, αλλά ακόμα αμφιταλαντεύονται, δεν υπάρχουν αλλαγέ σε σχέση με την κατάσταση που ίσχυε στι 3 Δεκάτου του 2014. Οπότε, η βελτίωση πρέπει να πούμε και να ομολογήσουμε είναι αρκετά περιορισμένη. Τώρα, ε, εμείς τι κάνουμε ε, σε σχέση με όλα αυτά. Αρχίσαμε να εκπονούμε μία μελέτη αντικτύπου. Το 2016 θα ολοκληρωθεί αυτό, έτσι, 15-16, για να κοιτάξουμε τις διάφορες επιλογές και δυνατότητες που έχουμε για να βελτιωθεί η προστασία των επιβατών των σιδηροδρόμων και να εξασφαλιστούν οι κανόνες παιχνιδιού ε, για τις σιδηρομικές επιχειρήσεις και μπορεί να αλλάξει ο κανονισμός σε κάποια στοιχεία. Αλλά μεταξύ αυτών θα πρέπει, μεταξύ άλλων δηλαδή, να μειωθούν οι εθνικές εξαιρέσεις. Τι σημαίνει αυτό να καταργηθούν οι εξαιρέσει για τις εχώριες υπηρεσίες και να περιοριστούν και άλλες εξαιρέσει γενικότερα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ ωραία. Έχετε να ρωτήσετε κάτι, να τοποθετηθείτε. Εγώ θέλω να πω κάτι. Αλλά εντάξει, εσείς να πέστε. Συγγνώμη κύριος Βαντεκάμπ. Αγγλικά, Ολλανδικά δεν έχει σημασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι συνέχεια δίνει, τι προτίθεται να κάνει. Θα τα δίνουν αυτά τα κράτη-μέλη, θα τα τιμωρήσουν, θα τα ενθαρρύνουν, τι θα τα κάνουν. Εγώ έχω μία παρεμφερή ερώτηση. Το 2007 όταν αποφασίσαμε, τότε βέβαια ε, υπήρχαν όχι εξαίρεσεις ακριβώς, αλλά ε, νόμιμες δυνατότητες ε, καθυστέρησης. Κάθε πέντε χρόνια, αν είχε κανείς ε, λόγους, μπορούσε να επιβάλει αναστολή. Άρα δηλαδή ε, με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε κανείς ε, να ξεκονομήσει χρόνο για την νομοθεσία. Αυτό όμως δεν γίνεται. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι τα, χρόνια, τα κράτη βέβαια που το έκανα αυτό κάθε πέντε χρόνια πρέπει να το αιτιολογούν. Τα γνωρίζετε τα κράτη, τα ελέγξατε ή απλά τα δέχεστε. Και μου κάνει εντύπωση και το εξή. Η Γερμανία δεν αναφέρεται πουθενά. Ξέρω όμω ότι στα δύο χρόνια ήταν απαραίτητο να αποφασίσει η Γερμανική Βουλή. Και εγώ τότε διαμαρτυρήθηκα. Ε, η Υπουργό Δικαιοσύνη το είχε παρουσιάσει το θέμα και κουβέντα δεν είπε ότι υπήρχε κάποια πρόβλεψη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο την Επιτροπή και το παρουσίασε σαν να ήταν δική της πρόταση. Όταν όμως από την αντιπολίτευση ελέγχθη ότι θα μπορούσε να δοθεί πιο οξύς τόνος, είπε αυτό απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δηλαδή προέκυψε πάλι η ίδια εικόνα. Ό,τι είναι καλό σε εθνικό επίπεδο το κάνω εγώ και για τα κακά φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θέλω λοιπόν πολύ συγκεκριμένα να γνωρίζω ε, συγγνώμη γιατί είμαι Γερμανός και ασχολήθηκα με αυτό, να μου πείτε σε ποιο σημείο η Γερμανία δεν εφάρμοσε και ίσως μπορείτε να μας πείτε και σε άλλες χώρες που δεν εφαρμόστηκαν αυτά που αποφασίστηκαν και αυτό που είπε ο κύριος Βίμ Βαντεκάμπ. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Τελικά η Κομισιόν τι κάνει όταν νόμοι του οποίου έχει θεσπίσει δεν εφαρμόζονται. Δεν νομίζω ότι είστε, μπορείτε να είστε ικανοποιημένοι με αυτό. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κοιτάξτε, με παρακάλεσε ο συνάδελφό μου να απαντήσω. Λοιπόν, να σας πω καταρχήν ότι όσον αφορά τις εξαιρέσεις, οι εξαιρέσεις είναι μια δυνατότητα μέσα στον κανονισμό. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη έχουν σαφώς τη δυνατότητα να εφαρμόζουν νόμιμα αυτές τις εξαιρέσεις. Γι' αυτό υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, έτσι ώστε κράτη-μέλη που έχουν δυσκολίες να εφαρμόζουν τον κανονισμό σε όλες τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες, σιγά σιγά να εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη τις οδηγίες αυτές. Και δεν χρειάζεται να αιτιολογήσουν για ποιο λόγο εξαιρούν κάποιες υπηρεσίες από την πλήρη εφαρμογή του κανονισμού. Το 2012 προβήκαμε σε αξιολόγηση και εκεί διαπιστώθηκε ότι εξαιρούνται κυρίως εκείνα τα άρθρα του κανονισμού που προκαλούν υψηλό κόστος. Ας πούμε, αποζημιώσεις, ε, παροχή βοήθειας για άτομα με αναπηρία ή επίσης οι προκαταβολές ε, σε περίπτωση ασφάλειας ή ασφάλισης. Πάντω αυτά είναι εξαιρέσει και σα λέω ότι τα κράτη-μέλη δεν υποχρεώνονται να αιτιολογήσουν. Πρέπει μόνο να πούν ε, κατά πόσον θα παρατείνουν αυτέ τις ε, εξαιρέσει ή όχι. Και στην περίπτωση όπου μιλάμε για υπηρεσίε μεγάλη απόσταση, αυτό ε, πρέπει να το έχουν εισαγάγει μέχρι το 24. Στην περίπτωση της Γερμανίας, η Γερμανία Στη Γερμανία δεν εξαιρούνται μεγάλες αποστάσεις. Ο κανονισμός ισχύει για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες, αλλά η Γερμανία εξαίρεσε τις αστικές ε, και περιφερειακές και υποπεριφερειακές υπηρεσίες και για συγκεκριμένο ε, χρονικό διάστημα. Καλωσορίζω τον κύριο Σπάχ ε, Μπαχ, με συγχωρείτε, γιατί ε, μιλάγαμε τόση ώρα για την έκθεσή του ε, και χαίρομαι που ήρθε επιτέλους. Όταν έρχεται κανείς ε, τελευταίος κάνει και εντύπωση, λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, όσον αφορά τις περιφερειακές αστικές συγκοινωνίες, αυτή ήταν η συμβαστική πρόταση επί της οποίας αποφασίσαμε, είπαμε αρχικά η Κομισιόν και το Συμβούλιο το επιθυμούσαν αυτό, αυτή τη ρύθμιση, μόνο για τι διεθνεί μεταφορέ. Και εμεί στο Κοινοβούλιο είπαμε, όχι αυτό δεν το κάνουμε. Γιατί αυτό θα σήμαινε ότι αν πάμε από την κολονία ε, προ Βρυξέλλε και από τι Βρυξέλλε προ Άχεν, αν έχει δύο ώρε καθυστέρηση δεν παίρνω τίποτα, αν πάω όμω για τη Λέγη, τότε κάτι θα πάρω. Αυτέ λοιπόν οι συζητήσει ε, κράτησαν μέχρι τη νύχτα, τρει η ώρα, και η συμβαστική πρόταση ήταν ότι ισχύει για τις ε, σιδηροδρομικές συνδέσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι όμως για τις αστικές και τις προαστιακές ε, συνδέσεις. Για τις μεγάλες αποστάσεις ισχύει αυτό, ακόμα και αν πάω από το Αμβούργο στο Μόναχο. Ήταν λοιπόν ένα συμβιβασμό ε, και νομίζω με αυτή τη συμβαστική πρόταση ήμασταν όλοι ευχαριστημένοι. Τώρα, ε, το θέμα είναι ότι αυτό επιτεύχθηκε και στις ε, μεγάλες αποστάσεις, Άρα δηλαδή θα πρέπει να κάνετε μια διαφορετική αξιολόγηση. Βεβαίως και θα ήταν καλό αυτή η ρύθμιση να ισχύει για τις ε, κοντινές και αποφάσεις, τις μικρές αποστα... κοντινές αποστάσεις, τις μικρές αποστάσεις. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι από αυτού, παρακαλώ. Κοιτάξτε, όπως σας είπα, οι μεγάλες αποστάσεις μπορούν να εξαιρεθούν τρεις φορές επί πέντε χρόνια, κατά το μέγιστο μέχρι το 2024. Και εδώ δημοσιεύσαμε στην ιστοσελίδα μας ε, μια έτσι σφαιρική εικόνα όπου βλέπετε ποια κράτη-μέλη έχουν εξαιρέσει τις εσωτερικές ε, σειρονομικές γραμμές μεγάλων αποστάσεων. Εδώ δεν εντάσσεται η Γερμανία. Από Μόναχο προς Αμβούργο ισχύει ο κανονισμός. Αλλά ας πούμε στη Γαλλία δεν ίσχυε πέρυσι ε, και μόλις φέτος ήρθησαν αυτές οι εξαιρέσεις. Πρόεδρος, κύριε Μπαχ, Θέλετε κάτι να πείτε? Θέλετε να μιλήσετε? Όχι. Ε, μήπως να του πω εγώ τι είπαμε. Είδαμε ε, ε, μια ταινία και έπαιζες. Äh, Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και τους επένους και τα συγχαρητήρια. Αλλά ας σοβαρευτούμε τώρα. Είχα μια συνεδρία και στην Επιτροπή Απασχόλησης και ξέρεις πώς είναι και αυτά τα πράγματα. Σημαντικές και καλές οι μεταφορές και άγιες, αλλά και η απασχόληση και τα κοινωνικά έχουν τη σημασία τους. Ε, ήμουν δικαιολογημένος. Ε, Λοιπόν, τώρα συζητάμε για τους επιβάτες των σιδηροδρομικών μεταφορών. Διάβασα την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την έκθεσή της. είχα ε, κάποιες σκέψεις και εγώ τότε και συμφωνώ με την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν με ικανοποιούν αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, καταγράφει πάρα πολλά προβλήματα, ε, τα οποία εγώ γνωρίζω και συναντάω καθημερινά. Δηλαδή, πραγματικά κυριαρχεί, βασιλεύει εκεί η ζούγκλα σε ό,τι αφορά ε, τα δικαιώματα των επιβατών. Υπάρχουν τόσες πολλές εθνικές ερμηνείες με τόσες εξαιρέσεις που πραγματικό εγώ θαυμάζω εκείνους που έχουν και μια συνολική εικόνα για όλα αυτά. Εγώ δεν μπορώ να εξηγήσω πολύ συχνά σε ένα πολίτη ε, τι δικαιώματα έχει και που μπορεί να διεκδικήσει το δίκιο του στο κάτω-κάτω. Και σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ερωτώ λοιπόν τώρα... Τι μέλη γενέστε, ναι, από εδώ και μπρο τι προτίθεστε να κάνετε. Δεν μπορούμε να καθίσουμε με σταυρωμένα τα χέρια να παρακολουθούμε τι συμβαίνει. Πρέπει να αναλάβουμε κάποια δράση. Εντάξει, ε, ε, λαμβάνουμε γνώση και υπόψη της αποφάσεις ε, των κρατών, αλλά καλό θα ήταν να τι καλέσουμε να δράσουν. Γιατί δεν διαφαίνεται και καμιά αλλαγή για κανένα τέλος αυτή την κατάσταση. Τα κράτη-μέλη ζητούν όλο και περισσότερες εξαιρέσεις και έχουν καθυστερήσει κιόλα πάρα πολύ ε, να ειδοποιούν και να ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι κι αλλιώς. Οπότε πρέπει από κοινού κάτι να κάνουμε, να αναλάβουμε δράση. Και ρωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι προτίθεστε να κάνετε. Εκτός από ε, αυτό τον απολογισμό που κάνετε, ε, τι μέλη γενέστε, θα αναλάβετε νέες πρωτοβουλίες, δεν το θεωρείτε σκόπιμο αυτό. Τι προτίθεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μία δεύτερη ερώτηση. Πριν από λίγους μήνες, εδώ στο Βέλγιο κυρίως είχαμε αυτή τη συζήτηση, το οποίο Βέλγιο ήταν πολύ επιφυλακτικό με τη χρήση των εξαιρέσεων, δηλαδή δεν έκανε χρήση πολύ. Και τώρα προτίθεται να εφαρμόσει πλήρως τις προτάσεις. Και εγώ φοβούμαι ότι οι χώρες που κινούνται ή που έχουν κινηθεί και τα έχουν όλα εφαρμόσει, τελικά είναι τα κορόιδα, για να το πω έτσι κάπως χοντρά. Ε, αυτά κατά την άποψή μου είναι απαράδεκτα πράγματα και θα πρέπει από κοινού να αντιδράσουμε. Ε, ε, τι προτίθεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γνωρίζει αυτές τις πρακτικές και τι προτίθεται να αναλάβει ως δράση σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Βεβαίω, δεχόμαστε τη συγγνώμη, είναι πολύ σημαντικέ οι συνεδριάσει των σκιωδών και χαιρόμαστε που τα κατάφερε και ήρθε Με ενδιαφέρει και με αυτό. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη Γερμανία υπάρχει μια παροιμία που λέει ότι όταν είσαι ειλικρινή δεν πρέπει να είσαι και κορόιδο και η έντιμη όμω τελικά αυτό αποδεικνύεται. Και άμα δεν εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό δίκαιο, τι να το κάνουμε. Μπορούμε και να το καταργήσουμε αν είναι άχρηστο το είχαμε σκεφτεί και εμείς και θέλουμε να κάνουμε και μια κριτική. Όταν έχουμε εξαιρέσει τρει φορές πενταετία μπορεί να υπάρχει μία-δύο χώρε που να έχει τεράστιο πρόβλημα. Αλλά δεν επιτρέπεται ποτέ να δίνουμε τέτοιες προθεσμίες και μάλιστα και αδικαιολόγητα να μπορούν να παρατείνουν και να ορίζουν τι πρόκειται να κάνουν, τι προτίθεται να κάνουν την επόμενη πενταετία και να είμαστε πολύ αυστηροί. Μετά όμως από αυτή την εμπειρία δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς δεν είμαστε, αλλά είμαι βέβαιος ότι και εσείς δεν είστε. Ερώτηση λοιπόν τώρα τι θα κάνετε. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αυτό είναι σαφέστατο. Πώς μπορεί κανείς να είναι ικανοποιημένος με τέτοια κατάσταση. Ακόμα και αν διαβάζοντας τα κείμενα, νομικά ας πούμε, τα κράτη-μέλη που έχουν κάνει χρήση των εξαιρέσεων είχαν το δικαίωμα να το κάνουν. Και ήταν δικαίωμά τους και χωρίς αιτιολόγηση και δικαιολόγηση. Δυστυχώς, αλλά αυτό λέει το κείμενο. Αρχίσαμε λοιπόν εμείς να δουλεύουμε. Γίνεται τώρα μελέτη αντικτύπου και ε, με βάση αυτή θα κατέλθει μία νομοθετική πρόταση για το θέμα των εξαιρέσεων. Είμαστε στο στάδιο ακόμα της μελέτης αντικτύπου. Οι εξαιρέσει λοιπόν ε, ε, πρέπει να επανεξεταστούν και ε, όπως και άλλα ζητήματα σε σχέση με τα δικαιώματα των επιβατών των συνδρομικών μεταφορών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Κατόπιν τούτου κλείνει αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Πάμε στο 16 που είναι τα διάφορα. Δεν υπάρχει τίποτα. Κατόπιν τούτου θα συναντηθούμε την, 12 ε, Οκτωβρίου, 3 η ώρα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ήσασταν πολύ αλλά ουσιαστικοί. Και μέχρι τότε να περνάτε καλά.